Mes συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Λίγη ησυχία παρακαλώ, διότι είναι πάρα πολύ φορτωμένη η ημερήσια, μας, η διάταξή μας για σήμερα το απόγευμα και γι' αυτό θα ήθελα να τηρούμε τις χρονοθυρίδες που έχουμε προβλέψει. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων. Αν σας φανώ απότομος ε, στη συνέχεια, έχετε δει την ημερήσια διάταξη. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια, μπορούμε να προχωρήσουμε. Κατόπιν, άλλες ανακοινώσεις του Προέδρου. Έχουμε διερμηνία από και προς όλες τις γλώσσες. Είναι δημόσια η συνεδρίαση η σημερινή, όπως και όλες εξάλλου, και αναμεταδίδεται παγκοσμίω στο διαδίκτυο. Ε, έχουμε την ακρόαση πολυεθνικών εταιριών σήμερα, εταιριών που έχουμε προσκαλέσει για σήμερα. Πρωτού ξεκινήσουμε με την τραγωδία που έγινε στο Παρίσι πριν από λίγες μέρες θα ήθελα να σας ζητήσω να συμμετάσχουμε και εμείς στο θρήνο των οικογενειών με ένα λεπτό σιγής θυμούμενοι και θύματα ε, και άλλων επιθέσεων στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ. Ένα λεπτό σιγής παρακαλώ. Je vous remercie. Έχουμε προβλέψει λοιπόν την ακρόαση εκπροσώπων 11 πολυεθνικών εταιριών. Είδατε πως ε, επειδή έχουμε πέντε ώρες στη διάθεσή μας μέχρι τις 8 το βράδυ, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε αυστηροί ως προς τα οργανωτικά. Προβλέπετε λοιπόν πως θα έχουμε δύο πάνελ. Πέντε εταιρείε στο πρώτο πάνελ. Κατόπιν ερωτήσεις από τρεις ε, πολιτικές ομάδες, εκπροσώπους δηλαδή τριών πολιτικών ομάδων και άλλο ένα πάνελ με πέντε εταιρείες. Κάθε εκπρόσωπος εταιρείας θα έχει τη δυνατότητα να κάνει μια πεντάλεπτη εισαγωγική παρουσίαση. Στη συνέχεια, κάθε μέλος επιτροπής που έχει γραφεί στον κατάλογο θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ερωτήσεις για δύο λεπτά και έχουν πάλι στη διάθεσή τους πέντε λεπτά για τις απαντήσεις οι εκπρόσωποι των εταιριών. Η προσωρινή Επιτροπή Τάξ με την τωρινή της εντολή κάνει σήμερα την τελευταία της συνεδρίαση. Θα υποβάλουμε τα συμπεράσματά μας στις 25 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια και επιλέξαμε αυτήν την σημερινή ημερομηνία για να επιτρέψουμε στα μέλη της Επιτροπής να λάβουν υπόψη αυτά τα συμπεράσματα και να τα ενσωματώσουν στο σχέδιο έκθεσης που θα υποβάλουμε την επόμενη έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ηγεσία και τους εκπροσώπους των εταιριών για τη σημερινή τους παρουσία που επιβεβαιώνει ότι κανένας οικονομικός φορέας όσο πανίσχυρες και αν είναι οι πολυεθνικές εταιρείες δεν μπορεί να αρνηθεί να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά αυτό μας ικανοποιεί ιδιαιτέρως. Για τους προσκεκλημένους, ε, καθώς ε, και το ακροατήριό μας στην αίθουσα ή ε, μέσω του διαδικτύου, θα ήθελα να κάνω τις εξής διευκρινήσεις. Συγκροτήθηκε αυτή η προσωρινή επιτροπή μετά τις αποκαλύψεις του σκανδάλου Lux Leaks. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο μας έδωσε τότε την εντολή για μια εξεταστική επιτροπή για τις φορολογικές πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υποβάλουμε προτάσεις για να διορθώσουμε την κατάσταση σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΟΣΑ. Έχουμε ασχοληθεί ακριβώς με την εκπόνηση αυτών των συστάσεων από την αρχή του 2015. Δεν Έχουμε φορολογική αρμοδότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή δεν επιβαρύνει άμεσα τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Όμως ε, πρέπει εμείς να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον ε, προστατεύοντας σε βασικές αρχές όπως ε, ο θεμητός ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρείε, αλλά και τα κράτη-μέλη και ποιες είναι αυτές τις αρχές η διαφάνεια, η ισότητα, η δικαιοσύνη, ο ανταγωνισμός. Όμως ε, είδαμε ότι είναι ιδιαίτερα αδιαφανής και αθέμητος ε, ο ανταγωνισμός ε, και η διοχέτευση των κερδών από τις εταιρείες. Ε, διάφοροι όμιλοι, διάφορες εταιρείες έχουν εξαιτία αυτής της κατάστασης καταφέρει να πλουτίσουν εις βάρος άλλων και έχει παρέλθει πλέον αυτή η περίοδος για μας. Θα πρέπει η ζούγκλα αυτή να αντακατασταθεί από μια κατάσταση υγιούς και θεμητού ανταγωνισμού. Όπως για τις τράπεζες υπάρχει η κατάσταση πριν και μετά τους Lehman Brothers. Ε, έτσι λοιπόν μετά και πριν και μετά το Lex Leaks η κατάσταση δεν θα είναι η ίδια. Είδατε τα πορίσματα της Επιτροπής μας. Ε, δεν είμαστε ούτε ανακριτές, ε, ούτε δικαστές, ούτε εισαγγελείς. Ανήκουμε στο νομοθετικό σώμα και παρακολουθούμε τις έκνομες πρακτικές για να κάνουμε συστάσεις ούτως ώστε να αντικατασταθούν από ορθές πρακτικές. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω την εξής σύσταση. Ας αφήσουμε τα παραμύθια της χαλιμάς. Ξέρετε ότι ξέρουμε. Γνωρίζουμε ε, όλα τα έγγραφα που μας έχετε υποβάλει καθώς και τις ακροάσεις που έχουν κάνει εθνικά κοινοβούλια που έκαναν αντίστοιχες ακροάσεις στο παρελθόν ε, διάφορα άρθρα του ειδικευμένου τύπου. Έχουμε κάνει έρευνα σε ε, έξι περίπου χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελβετία. Έχουμε ως εκ τούτου ένα επίπεδο ενημέρωσης σχετικά υψηλό σε σχέση με τις τρέχουσες πρακτικές. Αυτό που μας ενδιαφέρει από την παρελθούσα και τωρινή σας εμπειρία είναι η φορολογική στρατηγική ευρωπαϊκή και παγκόσμια των ομίλων σας ε, δεδομένης και της τρέχουσας φορολογικής πρακτής. Θέλουμε να καταλάβουμε δηλαδή το εξή. σε πώς είναι δυνατόν το τωρινό φορολογικό πλαίσιο ενθαρρύνει τις ε, εταιρείε που βρίσκονται στην κορυφή ε, της κλίμακας να επιδίδονται σε αυτή την φορολογική δημιουργικότητα και θα θέλαμε να επεξεργαστούμε ιδέες για το βέλτιστο δυνατό φορολογικό πλαίσιο για την οικονομία του 21ου αιώνα. Και εξάλλου έχουν έρθει σε επαφή μαζί σας ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και του και ε, για τα κέρδη των εταιριών και η στρατηγική που αποκολουθείτε έχει εκπονηθεί πριν από έναν αιώνα. Έχει αλλάξει ο κόσμος, δεν υπήρχαν πολυεθνικές τότε, δεν υπήρχε η ψηφιακή οικονομία. Ποιο είναι το σύστημα, ποιοι είναι οι κοινοί κανόνες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο θα μας επέτρεπε να οδηγηθούμε σε διαφανέστερο, σε θεμητότερο ανταγωνισμό για να μπορέσετε κι εσείς ε, να ασχοληθείτε με τις επαγγελματικέ δραστηριότητες και να αποκομίσετε το προσδοκόμενο κέρδος, αλλά από πλευρά μας να ε, ε, έχουμε κι εμείς τη δυνατότητα με ισότιμους όρους ανταγωνισμού, κυρίως φορολογικού ανταγωνισμού, να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες κατόπιν. Ε, σε διάφορα κράτη-μέλη ή σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βάσει του διαχωρισμού των εξουσιών όταν υπάρχει υπόθεση ενώπιον της δικαιοσύνης θα απόσκουμε. Έχετε λοιπόν τη διακριτική ευχέρεια ε, σε, αυτή την περίπτωση να μην απαντήσετε σε ερωτήματα που ενδεχομένως ε, τεθούν. Αυτά εν είδη εισαγωγής και θα περάσουμε στο πρώτο πάνελ. Θα δώσω το λόγο στον Νίκλας Λούντμπλαντ ε, που είναι αρμόδιος για τις δημόσιες σχέσεις ε, στο Google, 5, στη Google. Πέντε λεπτά. Mr. Chairman, members of the committee, thank you for... Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκλωσή σας, περιμένω τις ερωτήσεις σας και χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνουμε κάποιες εισαγωγικές παρατήρησεις. Είναι η σωστή ώρα να δούμε πώς πληρώνουν φόρους οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Είναι στην επικαιρότητα το θέμα αυτό σε διάφορα μέρη όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία όπου συμμετέχουμε σε αντίστοιχες τέτοιου είδους συζητήσεις. Εμείς είμαστε ενός απλού αλλά και διαφανού συστήματος. Ο πρόεδρος μας έγραψε στους Financial Times εδώ και δύο χρόνια ότι απαιτείται ε, να ληφθούν υπόψη οι διαδικασίες όπως αυτή την οποία ξεκίνησε ο ΩΣΑ. Είπαμε επίσης ότι οι κυβερνήσεις είναι αυτές που θα καταθέτουν τους κανόνες και οι επιχειρήσεις θα υπακούουν. Εμείς προσπαθούμε στα πλαίσια της πληρωμής των φόρων της εταιρείας μας να σεβόμεθα τους κανόνες αυτούς. Χρησιμοποιούμε τις φορολογικές δομές όπως είναι γνωστές και χρησιμοποιούνται από πάρα πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις. Είμαστε μια παγκόσμια ε, επιχείρηση σε 40 χώρες Έχουμε εταίρους και συνεργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη έχουμε έδρα στην Ιρλανδία. Έχουμε 5.000 υπαλλήλου εκεί που εξυπηρετούν την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Έχουμε επενδύσει δισεκατομμύρια σε ευρωπαϊκές υποδομές και σε εταιρικέ συμφωνίες. Ε, παρά τις ε, επενδύσεις αυτές η Google όπως και άλλες ε, ε, μεγάλες επιχειρήσεις πληρώνουμε τους περισσότερους φόρους μας στη μητρική μας χώρα. Εμείς δώσαμε περίπου 3,3 δις. Το 88 δόθηκε στην Ομοσπονδιακή Αμερικανική Υπηρεσία Φορολογίας. Αυτό οφείλεται στο ότι ο φόρος εισοδήματος βασίζεται στα κέρδη και όχι στα έσοδα ή την έδρα των πελατών της επιχείρησης και αυτό λαμβάνει υπόψη και το πνευματικό κεφάλαιο, την τεχνογνωσία και την τεχνολογία που βρίσκεται στη βάση της διεθνούς διαφημιστικής μας δραστηριότητας. Τα κόστη και οι κίνδυνοι της ανάπτυξης αυτού του πνευματικού κεφαλαίου από την, ε, από την επιχείρησή μας αναλαμβάνεται από την Ιρλανδική θηγατρική και φυσικά εκεί μπορεί να υπάρχουν και ζημίες. Αυτό σημαίνει για την Google ότι αναπτύσσουμε την τεχνολογία μας με κάποιο κόστος και αυτό δεν θα πρέπει να το υποτιμάτε. 9,2 δις δώσαμε στην έρευνα και τεχνολογία. Κάποιες από τις δαπάνες αυτές τις πλήρωσε η Google Ireland. Εμείς επιλέξαμε την Ιρλανδία για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων και το ελκυστικό φορολογικό περιβάλλον. Ε, υπήρξε μια συμφωνία με την Ιρλανδική κυβέρνηση, ε, όπως και με πολλές άλλες επιχειρήσεις οι οποίες πληρώνουν ακριβώς ε, με τον ίδιο τρόπο και στην Ιρλανδία και σε άλλες χώρες. Τώρα η δομή της φορολογικής μας αν θέλετε δραστηριότητας η Google Γερμανίας και η Google Σουηδίας όπου εργάζομαι καταρχάς ε, λειτουργούν σε επίπεδο εμπορικό. Ξέρετε ότι οι διαφαμιστικές συμφωνίες και συμβάσεις είναι περίπλοκες και πρέπει να ξοδεύουμε πάρα πολύ ε, χρήμα και χρόνο για να πείθουμε τις επιχειρήσεις να διαφημίζονται online. Έχουμε 300 σαν παράδειγμα ηλεκτρολόγους μηχανικούς οι οποίοι εργάζονται και για τις βαριές υποδομές στην Google Γερμανίας. Ε, προσπαθούμε να συνδυάσουμε, να αποφύγουμε επικαλύψεις. Ε, θα ήταν εναλλακτική βέβαια να προσφύγουμε σε εξωτερικούς εργολάβους για να καλύψουμε κάποιες από τις δραστηριότητες αυτές. Πάντως η δομή μας αυτή ακολουθεί αν θέλετε το σκελετό του συστήματος φορολογίας σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, στην Ιρλανδία σαν παράδειγμα έχουν αρχίσει βέβαια να αλλάζουν τα πράγματα, έχουν αρχίσει να γίνονται βήματα προόδου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κυβερνήσεις θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη φορολογική πολιτική για να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις. 26 από τις χώρες ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ε, δημιουργήσει κάποια κίνητρα για χρήση στον φορολογικό τομέα. Λυπάμαι λέει ο Πρόεδρος, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ε, αυστηροί και γι' αυτό προσπαθήστε να ισορροπήσετε κάπως την παρουσίαση της στρατηγικής σας και το τι σκοπεύετε να κάνετε στο μέλλον. Ε, στην εκπρόσωπο του Facebook τώρα είναι υπεύθυνη για τις δημόσιες πολιτικές της εταιρείας στη Νότια Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που δίνετε την δυνατότητα στη Facebook να εκφραστεί σήμερα. Είμαι υπεύθυνη της Facebook για την Νότια Ευρώπη, έχω έδρα στο Παρίσι που είναι και η έδρα του ΩΣΑ και παρακολουθώ τα θέματα της φορολογικής πολιτικής. Δεν είμαι ειδική στα φορολογικά, αλλά ελπίζω να αναφερθώ σε αυτά με επάρκεια. Το Facebook είναι μια αμερικανική επιχείρηση, η οποία λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρώπη έχει πολύ μεγάλη σημασία για το Facebook και ήρθα εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω τις επενδύσεις μας και τις δραστηριότητές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξηγήσω τη φορολογική μας δομή. Προσπαθούμε να καταστήσουμε τον κόσμο πιο ανοιχτό και διασυνδεδεμένο. Είμαστε καινοτόμος, ιδιαιτέρως καινοτόμος επιχείρηση και προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε στις νέες αλλαγές στον κόσμο. Έχουμε ένα δισεκατομμύριο, 600.000 εκατομμύρια πελάτες στον κόσμο, 315 εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι πελάτες μας. Ήδη από το 2008 οργανώσαμε τις δραστηριότητές μας με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο σε εμπορικό επίπεδο με τρόπο απλό και αποτελεσματικό σε επίπεδο χρηματοδοτικό. Να υπενθυμίσω ότι το πρότυπο το επιχειρηματικό μας συνίσταται στην πώληση διαφημιστικού χώρου online. Υπάρχει πολύ ισχυρός ανταγωνισμός, πολύ δυναμικός ανταγωνισμός. Λαμβανομένης υπόψη, ε, αν θέλετε, της δραστηριότητάς μας και του μεγέθους ε, του χώρου που καλύπτουμε, εμείς επενδύουμε ιδιαίτερο σε επίπεδο ε, προσωπικού και επίπεδο υποδομών. Είμαστε μια επιχείρηση παγκόσμια, αλλά είμαστε και μια ευρωπαϊκή επιχείρηση. Έχουμε 14 υπηρεσίες και θηγατρικές στην Ευρώπη με 1.700 υπαλλήλους. Η διεθνής μας έδρα είναι στο Δουβλίνο για την Ευρώπη, άνοιξε το 2009 και συνολικά 9.000 άτομα παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες στους πελάτες μας και στους χρήστες. Έχουμε στη διάθεσή μας και ένα κέντρο συλλογή στατιστικών στην Σουηδία. Ανοίξαμε φέτος ένα κέντρο έρευνας και τεχνητής νοημοσύνης στο Παρίσι. Έχουμε ε, μια υπηρεσία μελέτης και ανάπτυξης στο Λονδίνο και έχουμε και άλλα γραφεία στο Αμβούργο, στις Βρυξέλλες, στη Μαδρίτη, στη Στοκόλμη, στο Μιλάνο κτλ κάθε μέρα χρησιμοποιείται από τους ε, μικρομεσαίους επιχειρηματίες και νοτόμους δημιουργούς πνευματικού περιεχομένου που καλύπτουν όλο και περισσότερο και κίνο ε, και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας. Το δίκτυό μας ε, πάρα πολύ βασικοί εταίροι της νέας οικονομίας έχουν αναπτυχθεί όπως το Spotify και άλλες. Το 2014 Ε, ε, υπόθηκε ότι οι οικονομικές επιπτώσεις αν θέλετε ε, οι δραστηριότητες της επιχείρησής μας στην Ευρώπη φτάνει τα 51 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει ελπίζω να αναπτύσσεται. Είμαστε υπέρ του ενιαίου οικονομικού χώρου και νομίζω ότι αυτό θα ωφελήσει συνολικά την κοινωνία. Για να επανέλθω τώρα στην ουσία της συζήτησης, εμείς λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τις φορολογικές μας υποχρεώσεις. Πληρώνουμε αυτό το οποίο απαιτείται και στην Ευρώπη. Έχουμε θύγατρικές επιχειρήσεις στα πλαίσια μιας μητρικής που έχει έδρα την Ιρλανδία. Αυτό καλύπτει το σύνολο του κόσμου εκτός Βορείου Αμερικής. Ε, το μοντέλο το ε, έκανε την περιγραφή του και ο παρακαθήμενος προηγουμένως. Έχουμε διάφορες υπηρεσίες που στηρίζουν τις διεθνείς εμπορικές μας δραστηριότητες όπως το consulting στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, στις μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες. Έχουμε επίσης και άλλες θηγατρικές επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται περισσότερο με τη διαχείριση των κέντρων συγκέντρωσης δεδομένων όπως επίσης και της εξυπηρέτησης των χρηστών. Τώρα για τον τελειώνω Πέντε λεπτά, δεν έχω περισσότερο χρόνο και το λέω και για τους επομένους. Παρακαλώ, μην παρουσιάζετε τόσο την επιχείρησή σας γιατί την ξέρουμε την επιχείρηση και να περνάτε απευθείας στην ουσία, δηλαδή στο θέμα της φορολογίας των κερδών. Πώς ακριβώς βλέπετε την φορολογία των κερδών. Θα ξαναπάρετε το λόγο προηγουμένω και θα απαντήσετε στις ερωτήσεις των μελών. Για την Amazon τώρα η κυρία Μίτσι αντιπρόεδρος σε παγκόσμιο επίπεδο ε, της ε, Amazon. Λέγομαι Μονίκ Μέσ και είμαι αντιπρόεδρος της Amazon για θέματα διεθνούς πολιτικής και δίπλα μου είναι ο κύριος Ντίσμαν που είναι αντιπρόεδρος αρμόδιος για θέματα φορολογίας. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας να εμφανιστούμε ενώπιον σας για να συζητήσουμε θέματα φορολογίας. Με χαρά θα ε, συμβάλλουμε στο έργο της Επιτροπής σας και θα καταθέσουμε τις απόψεις μας και ιδίως για το σχέδιο BEPS του ΟΣΑ καθώς και την ενιαία φορολογική βάση εταιριών άλλη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς λειτουργούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1998 και έχουμε πάνω από 35.000 εργαζόμενους σε 50 περίπου τόπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος μας είναι ο καταναλωτής με πολλές μικρές και μεσές επιχειρήσεις και αυτά βεβαίως εμφανίζονται και στην ιστοσελίδα μας. Ε, είναι και δικό μας το όραμα μιας πλήρως ενωμένης ενίας αγοράς που να βασίζεται και να συμμορφώνεται με τους κανόνες και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ενία Αγορά αλλά και διεθνώς. Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, σαφήνεια και ασφάλεια και για τους κανόνες και για την εφαρμογή τους είναι εργαλεία κλειδιά. Και γι' αυτό είμαστε υπέρ της προτάσεως του ΟΣΑ και για να υπάρξει και διεθνή συνένεση βέβαια. Ευτυχώς έχει επιτευχθεί συνένεση σε πολλούς τομείς, κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό λόγω και του σύντομου χρονοδιαγράμματος και βεβαίως και λόγω των πολλών ενδιαφερομένων μερών, stakeholder. Έχουμε υπάρχει ανάγκη να βασιστούμε στη συνένεση αυτή, ώστε οι μεταρρυθμίσεις που θα συμφωνηθούν να εφαρμοστούν με τρόπο συνεκτικό και συνεπή. Είναι σε ισχυρή θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να οδηγήσει σε συντονισμό και στην Ευρώπη και διεθνώς. Και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για να επιτύχει τα επόμενα κρίσιμα βήματα. Και πρώτο, επαρκώς μεγάλος αριθμός χωρών θα πρέπει να μπουν στην πολυμερή συμφωνία του ΟΣΑ το 2016, ώστε το BEPS να εφαρμόζεται με συντονισμένη βάση. Δεύτερο, οι χώρες θα πρέπει να εφαρμόζουν και τις διατάξεις για την κατανομή ε, ε, κερδών και οφειλών. Βεβαίως, από καιρού καιρών έχουμε και εμείς ζημίες, ιδίως όταν κάνουμε μεγάλες επενδύσει. Οι κανόνε για την κατανομή θα πρέπει να βασίζονται σε κοινή βάση και να προβλέπουν οι χώρες αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να αποφεύγεται το αλπιτράζ. Ιδίως όταν παραπάνω από μία χώρες λαμβάνουν διαφορετικές θέσεις σχετικά με την κατανομή των ζημιών και των κερδών. Αυτά για την σωστή μεταχείριση και των καταναλωτών και των φορολογικών αρχών. Υποστηρίζουμε λοιπόν το έργο του ΟΣΑ. Εμείς συμφωνούμε με, τις, με τους στόχους της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κοινή φορολογική ε, βάση για τη φορολόγηση των εταιριών. Και επιθυμούμε και εμείς να μειωθεί η περιπλοκότητα και το κόστος εφαρμογής των κανόνων. Συμφωνούμε με τα σχόλια από πολλές ε, οργανώσεις επιχειρήσεων που λένε ότι δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί ορισμένα πράγματα εφόσον παραμείνουν τα υψηλά κόστη. Οποιαδήποτε πρόταση λοιπόν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και καταστάσει ζημιών, όσο και την κατανομή των κερδών. Και αυτό είναι σημαντικό για εταιρείε όπω η Amazon, η οποία κάνει επενδύσεις με πολύ μεγάλο κόστος, αλλά και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αρχίζουν να δουλεύουν και που έχουν συχνά στην αρχή ζημίες. Ένα τρόπος για να βελτιωθεί η πρόταση θα πρέπει να είναι και η υποχρεωτική δεσμευτική διαιτησία, το σχέδιο που προβλέπει και ο ΩΣΑ, έτσι ώστε να αποφευθεί η διπλή φορολόγηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχουν σαφέστερε θέσει μεταξύ των χωρών μελών. Και ιδίω για τι διαφορέ, για την επίλυση διαφορών δηλαδή, που είναι σημαντική και για το επενδυτικό κλίμα στην Ευρώπη. Άρα θέλουμε μια μεταρρύθμιση, φορολογική μεταρρύθμιση που να προβλέπει σαφείς και απλούστερους κανόνες και να εφαρμόζονται με τρόπο συνεπή και συνεκτικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε τώρα ε, δραστηριότητα, αν θέλετε, και περνούμε στον κύριο Μακίναν της HSBC, του Συλλόγου Τραπεζών δηλαδή, υπεύθυνο για θέματα ε, φορολόγησης. Και βλέπετε το χρονόμετρο πάνω στον τοίχο εκεί ψηλά. Μακίνουν από την HSBC. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που έρχομαι εδώ σήμερα για να εκπροσωπήσω την HSBC στην Επιτροπή σας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μιλήσω για το πώς προσεγγίσουμε τα τις φορολογικές μας υποθέσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρωταρχικό ερώτημα που θέσατε και για το οποίο θέλετε απάντηση. Ποια είναι η προσέγγιση μας. Πρέπει να πληρώσουμε ε, τα τους φόρους που μας αναλογούν ε, στις, ε, στα κράτη όπου φορολογούμαστε και φυσικά θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ισχύοντες ε, κανόνες και φυσικά οι κανόνες που εφαρμόζουμε στις επιχειρήσεις μας έχουν ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα κέρδη στις χώρες που πρέπει. Δεύτερον, οι τεχνικές επιθετικής φοροαποφυγής δεν ακολουθούνται από την εταιρεία μας. Στη συνέχεια έχουμε την προσέγγιση της διαφάνειας. Πιστεύουμε στη διαφάνεια, στις σχέσεις μας με τις φορολογικές αρχές και υποστηρίζουμε τις δημόσιες εκθέσεις χώρα που προκύπτουν από την οδηγία ε, CRD4. Ε, είμαστε μια τράπεζα, ένας ε, τραπεζικός όμιλος και πολύ μέτοχοι, το κοινό, εσείς, ε, θα θέλατε να μιλήσουμε για την υπόθεση Swiss Leaks. Ε, πριν από 7 χρόνια συνέβη αυτό στην HSBC και τότε αναγνωρίσαμε και εξακολουθούμε να το αναγνωρίζουμε ότι η κουλτούρα και οι φορολογικές πρακτικές της εταιρείας μας τότε ε, ήταν απαράδεκτες. Καλωσορίζουμε την εξέλιξη της νομοθεσίας ε, ΦΑΤΚΑ της ΕΙΠΑ και την ε, παγκόσμια εφαρμογή της, ε, καθώς και το σύστημα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που αναμένεται να αρχίσει να ισχύει σε λίγα χρόνια. Πιστεύουμε ότι με τη μεγαλύτερη διαφάνεια ε, θα βοηθηθούμε και εμείς και οι πελάτες μας για την ε, ιδιωτική τραπεζική τι έχουμε κάνει αλλάξαμε άρδιν τον τρόπο λειτουργίας ε, του ομίλου μας στην ιστοσελίδα μας εξηγούμε με ακρίβεια τι ακριβώς έχουμε αλλάξει, αλλά πραγματικά θεμελιωδώς έχουμε τροποποιήσει τις πρακτικές μας, στις συναλλαγές μας με τους πελάτες, σε όλες τις επιχειρήσεις σε όλες τις θηγατρικές μας. Όταν γνωρίζουμε ή υποπτευόμαστε τους πελάτες μας ότι ε, προσπαθούν να ε, φοροδιαφύγουν ε, περνούν από τον έλεγχο που έχουμε προβλέψει και καταθέτουμε τα απαιτούμενα στοιχεία στις φορολογικές αρχές και πάβουμε την σχέση τράπεζα πελάτη. Στις 4 Νοεμβρίου η Επιτροπή σας ε, ήδη ε, εκπώνησε πολύ καλές συστάσεις μέσα στην έκθεσή της. Ε, τι εντοπίσαμε εμείς ακριβώς. Η αρχή της συνέπειας είναι πάρα πολύ σημαντική. Όπως είπε και η συνάδελφος από την Amazon, έχει νόημα να επικρατήσει η διαφάνεια. Δεύτερον, θα πρέπει να φορολογούμαστε εκεί όπου συμβαίνει η επαγγελματική δραστηριότητα. Και σας είπα ότι αυτή την πρακτική την ακολουθεί ούτως ή άλλως πλέον η HSBC. Και η τρίτη αρχή της διαφάνειας ε, μας βρίσκει σύμφωνο σε σχέση δηλαδή με τις φορολογικές αρχές ε, δημοσιότητα των πληροφοριών σε σχέση με το πού πληρώνει κάποιος τους φόρους ανάλογα με το πού ε, διεξάγονται ε, οι δραστηριότητες. Και χάρη σε αυτή την διαφάνεια ε, και τη νομοθεσία ΦΑΤΚΑ και τα κοινά πρότυπα υποβολής αναφορών και αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια για τους πελάτες αλλά και γενικότερα για την κοινωνία. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ τον κύριο Διευθυντή. Αυτό που είπατε για τις εκθέσεις αναχώρα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως. Είναι μια αρχή η οποία εφαρμόζεται στην δραστηριότητά σας αλλά όχι σε άλλες δραστηριότητες και είναι ένα θέμα το οποίο θα προκαλέσει πάρα πολλές ερωτήσεις από πλευρά των μελών. Ο κύριος Χάμπαρτ για τα Barclays ο οποίος έχει θα έλεγα τι ίδιε αρμοδιότητες με εσά αλλά στην Τράπεζα Barclays. Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να πάρω το λόγο. Λέγομαι Μαρκ Χάμπαρντ και είμαι υπεύθυνο φορολογίας για την Barclays από το τέλος του 2013. Έχω εργαστεί στο θέμα αυτό εδώ και 20 χρόνια και τέτοιες πρωτοβουλίες που θέλουν να απλουστεύσουν τη φορολογία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι θετικές. Γι' αυτό ακριβώς χαίρομαι που είμαι εδώ για να μιλήσω για τα BEPS και την κοινή βάση επιχειρηματική βάση επιβολής να κάνω ορισμένα θα έλεγα σχόλια σχετικά με τις δραστηριότητές μας. Χρησιμοποιούμε 130.000 ε, εργαζομένους ε, κυρίως σε κάποιες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένε Πολιτείες και η Νότιος Αφρική. Οι τράπεζες της Barclays παρέχουν πολλές πιστοτικές υπηρεσίες, λιανικές υπηρεσίες, επιχειρηματική τραπεζική δραστηριότητα, πιστοτικές κάρτες και επενδύσεις. Πληρώσαμε 3,49 δις λίρες σε φόρους σε κέρδη τα οποία ξεπέρασαν τα 2,26 δις λοιπόν ουσιαστικά το ποσοστό φορολογίας μας πέρυσι ήταν 45%. Φυσικά πληρώνουμε περισσότερο στις χώρες που έχουμε τις μεγαλύτερες δραστηριότητες, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένε Πολιτείες και στην Νότια Αφρική, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, η Price Waterhouse πρόσφατα εξέτασε τις 100 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Barclays είναι ο, ο υψηλότερος φορολογούμενος στη χώρα αυτή. Έχουμε κάνει αρκετές αλλαγές στον τομέα αυτό και στη δομή της επιχείρησής μας τα τελευταία χρόνια και σε σχέση με το τι κάνουμε και σε σχέση με το πώς το κάνουμε. Έχουμε δημοσιεύσει το 2013 τις λεγόμενες φορολογικές μας αρχές Αυτές οι φορολογικές αρχές αφορούν κάθε αποφάση στον τομέα της φορολογίας τις οποίες λαμβάνω εγώ και κάθε δράση την οποία αναλαμβάνει η Barclays. Οποιοςδήποτε φορολογικός προγραμματισμός για μας ή για τις πελάτες μας θα πρέπει να στηρίζει γνήσιες εμπορικές δραστηριότητες, να είναι συμβατό ε, με τον νόμο και τον κώδικα πρακτικής, ε, να είναι φορολογικού φορολογική δραστηριότητα η οποία είναι αναμενόμενη από τις αρχές της κάθε χώρας και να είναι συμβατές και να φαίνεται ότι είναι συμβατές με τους στόχους και τις αξίες της επιχείρησής μας. Ένα θέμα το οποίο τίθεται και σας ενδιαφέρει πολύ εδώ στο Κοινοβούλιο είναι η φορολογική διαφάνεια και η προσπάθεια που γίνεται για αναφορά σε αναχώρα. Εμείς πήραμε την απόφαση να ξεπεράσουμε ε, τις απαιτήσεις της CRD και δημοσιεύσαμε ε, ένα κατάλογο των δραστηριοτήτων μας άνα χώρα που περιλαμβάνει λεπτομέρειες ε, για τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των εργαζομένων, τα κέρδη και το φόρο τον οποίο πληρώνουμε σε κάθε χώρα. Είμαι υπερήφανος ε, για τις βασικές αυτές αρχές λοιπόν τις οποίες αποδεικνύουμε ότι σεβόμεθα. Στο θέμα που συζητάμε σήμερα νομίζω ότι το BEPS του ΟΣΑ είναι μια καλή προσπάθεια. Έχει σημασία να υπάρχει εμπιστοσύνη του κοινού στο διεθνές φορολογικό σύστημα και ελπίζω ότι το BEPS θα το πετύχει αυτό. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετική επίσης και η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το CCCTB, την Κοινή Επιχειρηματική Βάση Επιβολής. Αυτό είναι κάτι που θα μειώσει ε, το κόστος το γραφειοκρατικό για τις επιχειρήσεις. Δυσκολίες θα υπάρξουν βέβαια. Αυτά τα θέματα ελπίζω λοιπόν να τα συζητήσουμε επί μακρόν. Σας ευχαριστώ που ακούσατε τις αγωγικέ μου παρατηρήσεις. Alors, après ces exposés introductifs, je vais la parole. Μετά τις αγωγικέ σας παρατηρήσεις θα δώσω το λόγο σε τέσσερα μέλη μας, ευρωβουλευτές δηλαδή, που προσωπούν τις τέσσερις πολυπληθέστερες σε δύναμη ε, πολιτικές ομάδες και πρώτα τον κύριο Μπάλτς για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης τις κυρίες και κυρίους που είστε σήμερα εδώ στην Επιτροπή Τάξη. Θα ήθελα να είχατε έρθει από την πρώτη πρόσκληση που σας απευθύναμε αλλά δεν μπορώ παρά να θυμίσω κάτι που είχε πει ο Κόντραντ Άντεναουερ, ότι ο καθένας πρέπει να έχει το δικαίωμα να γίνεται λίγο εξυπνότερος κάθε μέρα. Ελπίζω λοιπόν ότι στο μεταξύ γίνατε λίγο εξυπνότεροι. Πάντως χαίρομαι που είστε εδώ. Τρία θέματα. Πρώτο. Πρέπει να αποκατασταθεί ένας έντιμος φορολογικός ανταγωνισμός στην Ευρώπη. Η Επιτροπή μας, και νομίζω μπορούμε να το πούμε αυτό, στάθηκε κριτική απέναντι στο ότι πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις διαρρυθμίζουν έτσι τις ε, διεθνείς τους δραστηριότητες ώστε να μπορούν να καταφεύγουν σε φοροαποφυγή. Και τελικώς μικρές και μεσές επιχειρήσεις πληρώνουν μεγαλύτερους αναλογικά φόρους. Πρώτη ερώτηση λοιπόν. Πώς βλέπετε τα φορολογικά σας πλονεκτήματα απέναντι στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις και ως μάνατζερ μιας μικρής επιχειρήσεως θα είχατε τις ίδιες επιλογές των οποίων χαίρουν τώρα οι επιχειρήσεις σας. Δεύτερο, θα ήθελα να μάθω λίγο περισσότερα πράγματα σχετικά με τον φορολογικό σχεδιασμό σας. Ποια εσωτερικά τμήματα έχετε στις επιχειρήσεις σας, δεν αναφερθήκατε όλοι σε αυτό τα οποία κάνουν τον φορολογικό σχεδιασμό. Και τρίτο, ποια είναι η ιεραρχία στο φορολογικό σχεδιασμό. Έχουμε δύο υπευθύνους από τράπεζες. Από τις άλλες επιχειρήσεις όμως υπάρχουν πλήθος ε, υπευθύνων για ε, φορολογικά θέματα. Ευχαριστώ κύριε Βάλτς. Ο ε, Πέτερ Σίμων, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε από σοσιαλδημοκρατική σκοπιά σωστό είναι να πω και εγώ ορισμένα πράγματα για το μέχρι τώρα ιστορικό της Επιτροπής. Σημειώσαμε ότι δεν δεχθήκατε την πρώτη μας πρόσκληση, την οποία εμείς θεωρήσαμε ως περιφρόνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη στάση σας αυτή δηλαδή. Για την σημερινή πρόσκληση βέβαια το ξανασκεφτήκατε και σας προτρέπω θερμά το ίδιο να κάνετε και σε μελλοντικέ προσκλήσεις, δημοκρατικά όργανα, δημοκρατικά εκλεγμένων κοινοβουλίων έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν και ποινικέ κυρώσει, Εννοώ εθνικά κοινοβούλια. Εμεί δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα. Να είστε όμω βέβαιες και βέβαιοι ότι έχουμε άλλα εργαλεία, έχουμε άλλα βέλη στη φαρέτρα μα, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον για να ε, επιβάλλουμε την βούλησή μα. Τώρα πιο συγκεκριμένα στι ερωτήσει μου. Πρώτα, για την Google το 2012 εξ όσων γνωρίζω, πληρώσατε 8,8 δισεκατομμύρια για την χρήση αδειών. Μιλήσατε επίσης πριν από λίγο για επενδύσεις στην έρευνα στην Ιρλανδία. Θεωρώ ότι στην ίδια τη Βερμούδ, στις ίδιες Βερμούδες δεν ε, κάνετε τόσο πολλές έρευνες και όμως πληρώνετε άδειες για χρήση ευρεσιτεχνιών. Πώς θα μου το εξηγήσετε αυτό, ότι η έρευνα δηλαδή γίνεται στην άλλη άκρη του κόσμου, όμως οι άδειε για τη χρήση των ευρεσιτεχνιών γίνονται, πληρώνονται από εσά σε άλλο τόπο. Και τελικώς αποφεύγετε να πληρώσετε πρόσθετε φόρους. Παρόμοια ερώτηση έχω για την Amazon. Πώς θα εξηγήσετε στους πολίτες ότι χρησιμοποιείτε, εποφελείστε από τις σύγχρονες υποδομέ πολλών χωρών μελών για την διακίνηση των εμπορευμάτων σας δεν πληρώνουν το φόρους. Το 2015 πληρώσατε παραπάνω στο Ενωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία και στην Ισπανία, αλλά ποια είναι ακριβώς η εικόνα και τι γίνεται σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα Γαλλία και Πολωνία. Θα πράξετε εκεί τα ίδια. Μάλιστα, σα ευχαριστώ αγαπητέ. Ο κύριος Λούκε, Μπέντ Λούκε, εξ ονόματος των ε, Ευρωπαίων Μεταρρυθμιστών και Συντηρητικών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ερώτηση προς την εκπρόσωπο της εταιρείας Facebook. Παρουσιάσατε την επιχείρησή σας, δεν είπατε όμως πολλά για τα προβλήματα που αποτελούν το αντικείμενο των εργασιών της Επιτροπής μας. Ενώ άλλοι από εσά του προσκεκλημένου είπαν πιο συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω τώρα ποια είναι η θέση σας απέναντι στην πρόταση για μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις. Και πιο συγκεκριμένα για το γεγονός ότι το βασικό στοιχείο είναι αυτό το ενοποιημένο. Υποστηρίζεται την πρόταση αυτή ή θεωρείτε ότι ενδεχομένως εμπεριέχει μειονεκτήματα για την επιχείρησή σας. Και για να το πω πιο συγκεκριμένα, σας ερωτώ σχετικά με την φορολογική κατανομή που διαπιστώνει κανείς, παρατηρεί κανείς στην επιχείρησή σας. Στο Ενωμένο Βασίλειο το 2014 πληρώσατε, σύμφωνα με τα όσα λέει ο τύπος, 4.000 λίρες στερλίνες. Ενώ ο κύκλος εργασιών σας ήταν περίπου της τάξης των 100 εκατομμυρίων λιρών. Και συνολικά βέβαια βρίσκεται... Δεν θυμάμαι αν είναι τώρα δολάρια ή ε, στερινής, πάντως πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Προφανώς η ε στερηνες παντως προκειται για ενα παρα φόρων στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε μια προφανή ανισομέρεια, προφανή ε, δυσαναλογία. Από την άλλη μεριά πληρώνεται φόρους και στα νησιά Καϊμάν, όπου εκεί πληρώνεται και για την χρήση τελών, πληρώνεται τέλη για τις ε, ε, ευρεσιτεχνίες κλπ. Η ίδια ερώτηση λοιπόν που έκανε και ο κύριος Σίμων προηγουμένως. Πώς το εξηγείτε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Για λογαριασμό τώρα των φιλελευθέρων, ο κύριος Τόιρερ που ήταν και συνεισηγητής της εκθέσεως. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πρώτον, ήταν καιρός πραγματικά να προσέλθετε εδώ ενώπιον της ε, Επιτροπής Τάξε. Πράγματι, η πρόσκληση που σας απευθύναμε και που δεν δεχθήκατε αποτελεί περιφρόνηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, ερώτηση για την εταιρεία Google. Στην Βουλή των Κοινοτήτων, στη Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων, κάποιος εκπροσωπός σας δέχτηκε ότι η Google έχει θηγατρική επιχείρηση στις Βερμούδες για να υπερασπίζεται την διανοητική ιδιοκτησία του Google εκτός Ενωμένων Πολιτειών. Μόνο εκεί μπορεί να γίνει αυτό, γιατί δεν μπορεί να γίνει στις Ηνωμένε Πολιτείες ή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προστασία αυτή δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να γίνει εκεί. Τώρα, για Emerson, το 2015 δηλώσατε ότι θα πληρώσετε φόρους στη Μεγάλη Βρετανία και στην Γερμανία. Γιατί ξαφνικά από Σαούλ γίνατε Παύλος. Προς άλλους τώρα εκπροσώπους. Χρησιμοποιείτε ευρεστεχνίες στην ε, Ολλανδία, στην Ιρλανδία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο και ποια είναι τα πλανεκτήματα, ποια είναι τα ε, ωφελήματα που λαμβάνετε από αυτά. Έχετε θυγατρικές σε νησιά Καϊμάν, Βερμούδες, τα κτλ. Και τέλος, για αυτή την βελτιστοποίηση των φόρων που στην ακρόαση της Βουλής των Κοινοτήτων επιβάλλεται στις ε, πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ποιος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, οι χώρες των ευρών των επιχειρήσεων αυτών ή τις συστάσεις αυτές τις γράφουν και δημοσιεύουν τα αρμόδια τμήματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, να ακούσουμε τις απαντήσεις. Ίσως με την ίδια σειρά, αν θέλετε. Κύριε Μπλαντ, ε, ακούσατε ερωτήσεις ειδικά για, την, ε, για τον όμιλό σας Google. Πέντε λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να εξηγήσω την κατάσταση, διότι είναι καυτό το ζήτημα και υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα. Λοιπόν, ε, το holding που έχουμε στην Ιρλανδία έχει έδρα στις Βερμούδες και για τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε μια εταιρεία που έχει την έδρα της στην Ιρλανδία και συναλλάσσεται με άλλες χώρες και άλλες περιοχές του κόσμου ε, έχουν ε, καταβληθεί φόροι στην Ιρλανδία και Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι ολόκληρη η δομή στις ε, Βερμούδες δεν διαγράφει ε, οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση, απλώς καταλογίζονται διαφορετικά φόροι που έπρεπε να έχουν καταβληθεί στις ΗΠΑ. Ε, Τώρα ε, εξετάζεται μεταρρύθμιση του συστήματος ε, και όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να είναι πιο προβλέψιμο και διαφανέστερο το σύστημα και παρακολουθούμε την διαδικασία και φυσικά όταν τροποποιηθεί η νομοθεσία θα συμμορφωθούμε και εμείς με αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σημαντικό να ε, δούμε ότι ε, δεν έχει σχέση με φόρους που θα καταβάλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η δομή στις Βερμούδες. Έχει σχέση με φόρους που κανονικά θα καταβάλλονταν στις Αμερικανικές αρχές. Κατόπιν μας ε, ρωτήσατε ποιες είναι οι οι σχέσει τη φορολογική στρατηγική και των φορολογικών αγώνων με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Υπάρχουν οι μικροπολιεθνικέ εταιρείε χρησιμοποιούν αντίστοιχα συστήματα με εμά και καταβάλουν φόρους για προϊόντα που πολλούν από την χώρα τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Εταιρείε με δημοφιλείς εφαρμογές, παραδείγματο χώρη, που ε, ε, καταβάλουν τους φόρους στη χώρα τους, ανεξαρτήτως που έχουν πουλήσει τις εφαρμογές στην Ασία, στην Αμερική κτλ. Ίδιο φορολογικό σύστημα, ίδια δομή για αυτές τις μικροπολιεθνικές εταιρείε ε, γιατί είναι εξίσου ε, επιτυχημένες όπως και οι παλιές ε, παραδοσιακές πολυεθνικές. Όπως όλες οι πολυεθνικές εταιρείες, αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται τελικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Υπάρχουν διάφοροι σύμβουλοι ε, και τους εξηγούν τι μπορούν να κάνουν σε σχέση με, την, ε, με το νόμο και με την νομοθεσία με την οποία πρέπει να συμμορφωθούν, αλλά η απόφαση παίρνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ε, Πάντω και στο άλλο σας ερώτημα έτσι. Αυτές τις ερωτήσεις είχα σημειώσει, νομίζω. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πρόεδρος, αν κατάλαβα καλά, μας είπατε πως η χρήση του double Irish μπορεί να συνδυαστεί με το Ολλανδικό σάντουιτς και να έχει ως αποτέλεσμα να αναβάλλεται η καταβολή φόρου και τελικά να διαγραφούν φόροι που έπρεπε να κατευθυνούν στις Αμερικανικές αρχές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αφορά αυτό φόρους ε, που έπρεπε να καταβληθούν σε ευρωπαϊκές χώρες. Ε, σωστά τα λέω. Απάντηση. Όχι, υπάρχει ε, αναβολή, όχι διαγραφή της φορολογικής υποχρέωσης, διαφορετικούς καταλογισμούς φορολογικών υποχρεώσεων. Ε, από τον Πρόεδρο θα μας βοηθούσε να μας το στείλει και γραπτός αυτό. Η κυρία Χέρ για το Facebook. Ναι, Πρόεδρε, θα προσπαθήσω γέρος να δώσω τις απαντήσεις. Δεν φτάνω το μικρόφωνο καλά-καλά, ελπίζω να με ακούτε καλά. Για τις ε, ερωτήσεις, για την Αγγλία, θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Είναι πολύ σημαντική η θηγατρική μας ε, στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε πλήρη ανάπτυξη. Απασχολούνται εκεί εξαιρετικοί εμπειρογνώμονες για το μάρκετινγκ και το προσωπικό μας ε, το αντλούμε από μια πολύ ανταγωνιστική αγορά ε, θα τα ξέρει ε, ο συνάδελφος από την Ελλαδία και δεν είναι, πολύ περιορισμένος αριθμός των ανθρώπων που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά και άρα πρέπει να δώσουμε γενναιόδορη αμοιβή κυρίως ε, να προσφέρουμε μετοχές σε αυτούς τους ανθρώπους για να τους προσελκύσουμε. η βάση μας ε, αυξήθηκε κατά 37% φέτος από το 2014 μέχρι ε, τώρα δηλαδή και ε, αυξήθηκε και ο ρυθμός των μετοχών και για συγκυριακούς λόγους υπάρχει μεγαλύτερη έκπτωση φόρου ως εκ λοιπόν ή, το 2014 ε, κατέβαλε περιορισμένους φόρους η θηγατρική μας ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αληθεύει αυτό. Κατόπιν μας κάνατε ερωτήσεις για την ενοποιημένη ε, βάση CCDTB. Ζητώ συγγνώμη, σχεδόν όρθια πρέπει να κάθομαι για να με ακούτε. τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις για να ξέρουν πώς να επενδύσουν και πώς να ε, αναπτυχθούν. Χρειάζεται προβλεψιμότητα και σταθερότητα των φορολογικών κανόνων. Στο μέτρο που είναι λειτουργικοί αυτοί οι κανόνες και προβλέψιμοι, οι καινοτόμες εταιρείε έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν. Η ενοποιημένη βάση είναι ένα μοντέλο που είναι συμβατό με τους δικούς μας στόχους, αλλά δεν είναι δική μας η απόφαση. Είναι αποφάσεις που λαμβάνουν σε εθνικό επίπεδο. Ε, οι που μας κάνει σε σχέση με τα νησιά Κάιμαν. Όπως και η Google, θα σας απαντήσω ότι έχουμε τις άδειες εκμετάλλευσης ε, ε, στα νησιά Κάιμαν, ε, αλλά ισχύουν διεθνώς, παγκοσμίως. Όταν λοιπόν υπάρχει ανάπτυξη παγκόσμιας ε, κλίμακας, εσείς αν μας μιλάτε για φορολογική δημιουργικότητα, εγώ θα μιλούσα για φορολογικό συντηρητισμό, διότι ε, είναι παραδοσιακές πλέον αυτές οι πρακτικές, ούτως ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί μια εταιρεία ε, σε παγκόσμια κλίμακα. Προσπάθησα να σου το εξηγήσω στην εισαγωγική μου παρουσίαση και γι' αυτό το λόγο τα πνευματικά μας δικαιώματα είναι ε, στα νησιά Καϊμάν. Το στιγμιότυπο το σημερινό για το ε, επιχειρησιακό μας μοντέλο είναι σημερινό θα μετεξελιχθεί για όλους τους λόγους που προανέφερα. Δεν είχα και πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες ε, του ΩΣΑ και ε, τη ομάδας εργασίας για τον ΠΕΠΣ, καθώς και ε, σε σχέση με την τροποποίηση της φορολογικής εταιρικής έδρας που έλαβε η Ιρλανδική κυβέρνηση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Δύο παρατηρήσεις να μου επιτρέψετε να κάνω. Καταρχάς μου κάνει εντύπωση όπως και ο προηγούμενος ομιλητής είπατε, ότι το ότι προσφεύγεται σε αυτό το οποίο ονομάζουμε κοινώς Double Irish με μια θηγατρική Ιρλανδική η οποία όμως έχει έδρασε ένα φορολογικό παράδεισο έχει συνέπειες στη φορολογία στη ΣΥΠΑ αλλά όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου κάνει εντύπωση, δεν προσκαλέσαμε την Apple σήμερα, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Όταν είχαμε πάει στις ΗΠΑ και επισκεφτήκαμε τον κύριο Tim Cook, τον γερουσιαστή που είχε ασχοληθεί με την Apple, και είδα τα πρακτικά της συνάντησής τους με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και είπε ότι χρησιμοποιεί την ρύθμιση τη φορολογική Double iris για να μην πληρώνει φόρο στην Ευρώπη αλλά να μην κλέβει καθόλου ε, τα φορολογικά έσοδα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Κοιτάξτε να διευκρινίσω κύριε Πρόεδρε. Το ότι η πνευματική ιδιοκτησία εδράζεται στα Κάιμανς δεν επηρεάζει την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών μελών αλλά την, ε, τη διαδικασία τη φορολογική στην Ιρλανδία. Αυτά για τις χώρες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Καλώς. Οπότε στην ουσία το πρόβλημα είναι ενδοευρωπαϊκό. Είναι ένα πρόβλημα ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο μας λέτε. Μία άλλη παρατήρηση την οποία αναφέρω κυρίως προς τους συναδέλφους μου. Ε, η περίπτωση του Facebook έχει ενδιαφέρον και θα ε, με ελέγχεται. Ε, η Facebook θεωρεί ότι η ανταγωνιστικότητά της, η δύναμή της βασίζεται στην ποιότητα φυσικά των ηλεκτρονικών ε, που χρησιμοποιεί, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό ακριβώς την οδηγεί να δίνει υψηλούς μισθούς, πολλά μπόνους, ε, μετοχές συγγνώμη, στους εργαζομένους, κάτι το οποίο μειώνει ε, ε, τα έσοδα τα, τα οποία πρέπει να φορολογηθούν. Νόμιμο είναι φυσικά αυτό. Έχετε κάτι να πείτε πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα να ανταπαντήσω. Έχει μεγάλη σημασία αυτό γιατί είναι το πρότυπο το οποίο ε, επιθυμούν να λειτουργούν οι καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Είναι μια συζήτηση αυτή η οποία έχει Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν τέθηκε το θέμα η συζήτηση για τα περιστέρια σε εισαγωγικά είναι ένα πρότυπο το οποίο θα χαρακτήριζα ιδιαίτερα χρήσιμο σε επίπεδο καινοτομίας ε, και αυτό οδηγεί και σε φορολογικές μειώσεις, διευκολύνσεις όπως και στη Γαλλία και είναι ένας μοχλός ουσιαστικά για την καινοτομία. Ο κύριος, ο Λου και πάλι. Μια σύντομη, εκεί είναι τα ακουστικά σας τα έχετε, ε, ε, σύντομη συμπληρωματική ερώτηση. Εάν κατάλαβα καλά, η διανοητική σας ιδιοκτησία έχει τοποθετηθεί στα νησιά Καϊμάν, ώστε το Facebook να μπορεί να αντιδρά γρήγορα και ευέλικτα. Γιατί άραγε δεν μπορεί να αντιδρά γρήγορα και ευέλικτα εάν προστατεύεται η διανοητική του ιδιοκτησία στην Γερμανία ή στη Γαλλία για παράδειγμα. Η απάντηση. Το μοντέλο που έχουμε διαλέξει είναι πολύ συντηρητικό και αυτό που χρησιμοποιείται συνήθως από επιχειρήσεις που δρούν στην αλλοδαπή. Και όταν βγήκαμε στο εξωτερικό, τέσσερα, χρονών είμαστε μόνο. Και έτσι λοιπόν ακολουθήσαμε το γενικά εφαρμοζόμενο μοντέλο που επιτρέπει να τοποθετήσει κανείς την προστασία της διανοητικής θεωρητικής σε κάποιο ουδέτερο τόπο που να επιτρέπει να ε, καλύπτει όλο τον κόσμο. Και όπως είπε και ο εκπρόσωπος του Google, η ιδιαιτερότητα είναι ότι στις ΗΠΑ, οι ΗΠΑ φορολογούν την διανοητική διοκτησία στο σύνολο του κόσμου και επομένως οι επιχειρήσεις ε, έχουν το κίνητρο να πάνε να εγκατασταθούν σε μια ουδέτερη τοποθεσία. Ε, μου άρεσε πράγματι αυτό το ουδέτερο που είπατε. Ο κύριος Λάμπερτ λέει, μα κοιτάξτε ένας τετράχρονος που ήδη δρά συντηρητικά. Δεν έχετε το λόγο, αγαπητέ φίλε. Πάντως μας άρεσε το αστείο. Ο κύριος Μακίναν. Α, με συγχωρείτε πρώτα, η κυρία Μέση. Να τα πει ο κύριος ε, Τίσμαν. Πρώτα, για τις πολιτικές μας για το φορολογικό. Εμεί περνάμε στο Amazon από τον Chief Financial Officer. Σύνηθες αυτό για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές, το πρώτο πράγμα που εξετάζουμε είναι να συμμορφούμαστε απόλυτα με τον ισχύοντα νόμο και με όποιο δίκαιο προβλέπουμε ότι θα εφαρμοστεί. Εάν πρόκειται να επέλθουν φορολογικές αλλαγές, επιθυμούμε να συμμορφωνόμαστε και με αυτές. Όσον αφορά τώρα το πώς προσεγγίζουμε την φορολογική εργασία, αυτές εξαρτώνται από τους καταναλωτές. Προσπαθούμε να υποστηρίζουμε δηλαδή τις πρακτικές των καταναλωτών. Για τη δεύτερη ερώτηση, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όντως πιστεύουμε ότι οι ίδιοι κανόνες πρέπει να ισχύουν για μεγάλες υποεθνικές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από την ιστοσελίδα μας πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων πολλούν τα προϊόντα τους και νομίζουμε ότι πρέπει να χαίρουν του ίδιου καθεστώτος. για τα διάφορα συστήματα και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τα συντονίσει. Ένα βασικό χαρακτηριστικό για τους επόμενους 18 μήνες θα είναι όσο περισσότερες χώρες δυνατόν να μπουν σε αυτό το πολυμερές εργαλείο εντός εισαγωγικών. Δύο χώρες όταν έχουν συνδιαλλαγές κάνουν μια συμφωνία, συνάπτουν μια συμφωνία μετά από διμερεί διαπραγματεύσει. Τώρα με το σύστημα BEPS, BEPS θα μπορεί να γίνει σε πολυμερή βάση και είναι σημαντικό να γίνει αυτό, να ε, γίνει δηλαδή να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό ε, ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού και αυτό είναι σημαντικό και για τους φορολογούμενους και για τις φορολογικές αρχές και από τις πιο βασικές προτεραιότητες κατά τη γνώμη μας. Να διασφαλιστεί δηλαδή ότι θα υπάρχει ε, ισότιμος ανταγωνισμός. Τώρα ακούστηκαν και άλλες ερωτήσεις, ε, φορολογικοί συντελεστές, κέρδη και άλλα σχετικά. Εμείς επενδύουμε σημαντικότατα στην Ευρώπη. Έχουμε και πάνω από 35.000 εργαζομένους στην Ευρώπη. Και τα κέρδη μας δεν είναι πάρα πολύ υψηλά. Είναι χαμηλό το ε, ποσοστό κέρδους μας. Μάλιστα είχαμε και ζημία το 2014. Βεβαίως, ότι, βεβαίως γνωρίζετε ότι οι φόροι επιβάλλονται επί των κερδών και όχι επί των εσόδων, όπως καμιά φορά λένε οι εφημερίδες. Η κυρία Μπρέσ. Σεβόμεθα πλήρως τις εργασίες της Επιτροπής σας. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η Επιτροπή σας. Δεν δεχθήκαμε τις προηγούμενες προσκλήσεις σας σε σχέση με τις ειδικές φορολογικέ ρυθμίσεις γιατί αυτή τη στιγμή υφιστάμεθα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα μια επίσημη έρευνα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεσμευόμεθα στα σχόλια τα οποία μπορούμε να κάνουμε σε θέματα φορολογικής πολιτικής. Σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σάιμον και ο κύριος Τόιρερ προηγουμένως. Στις αρχές του χρόνου εμείς ανοίξαμε ε, νέες επιχειρήσεις στην ε, Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό αποφασίστηκε πριν δύο χρόνια. Είναι μια απόφαση για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τις επιχειρήσεις μας αλλά και τους πελάτες μας φυσικά. Γι' αυτό ακριβώς και είστε υπέρ της έκθεσης αναχώρα. Γιατί ακριβώς έχετε δημιουργήσει θεατρικές επαφέ στις μεγαλύτερες από τις ευρωπαϊκές χώρες. Κοιτάξτε, θα το δούμε αυτό μιλώντας περισσότερο με τις φορολογικές αρχές και εξηγώντας τους τον τρόπο λειτουργίας της Amazon. Νομίζω ότι στην παρούσα φάση η εικόνα είναι επαρκής. Ο κύριος Μακίνεν. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν είχαμε έρθει νωρίτερα. Δεν είχαμε προλάβει να οργανωθούμε εδώ, αλλά ετοιμαστήκαμε και καταφέραμε να έρθουμε σήμερα. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν και έχουν σχέση με τις ψηφιακές επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο έχει σημασία νομίζω είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένες οι φορολογικές μας ομάδες, τα τμήματα και πώς εσείς έχετε την οργάνωση του ελέγχου για να βεβαιώνετε ότι πληρώνουν φόρους ή επιχειρήσεις αυτές. Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά να πούμε ότι στις περισσότερες οργανώσεις στις οποίες έχω πάρει μέρος πρέπει να ξεκινήσει κανείς τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στο Διευθυντικό Συμβούλιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο και από εκεί και πέρα να ελεγχτούν οι εφαρμογές, οι τρόποι εφαρμογής αυτών των αποφάσεων. Και αν πραγματικά δεν λαμβάνονται αποφάσεις για τη φορολογία σε επίπεδο διευθυντικό, τα προβλήματα είναι σοβαρά. Αλλά εφόσον ληφθούν οι αποφάσεις για τη φορολογία σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, τότε από εκεί και πέρα αυτό το οποίο έχει σημασία όταν τεθεί ένα φορολογικό θέμα είναι να είναι ξεκάθαρο το ποιος είναι υπόλογος και υπεύθυνος. Έγιναν και κάποιες άλλες ερωτήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να προσθέσω κάτι ουσιώδες εδώ. Σας ευχαριστώ. Ο επόμενος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. για τα τμήματα που ασχολούνται με τα φορολογικά, για τις διευκολύνσεις τις φορολογικές απέναντι στις μεγάλες επιχειρήσεις και την έλλειψη αντιστοίχων για τις μικρομεσαίες. Νομίζω ότι οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο. Οι μεγάλες επιχειρήσεις εργάζονται σε πολλές χώρες. Εμείς σαν πάκλε, σε 50 χώρες και αυτό δημιουργεί κάποια περιπλοκότητα. Και μπορεί να δημιουργεί προϋποθέσεις ε, για φορολογικές διευκολύνσεις, αλλά μπορεί να δημιουργεί και κινδύνους για φορολογικές ε, διπλές, για διπλή φορολογία. Πάντως στα πλαίσια του BEPS ε το θέμα είναι σωστό να επιδιώκεται να πληρώνονται οι φόροι εκεί όπου αναλαμβάνονται οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι και διεξάγεται η δραστηριότητα. Αυτό αντικατοπτρίζει τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα στο Barclays όταν προγραμματίζουμε τα θέματα τα φορολογικά, όπως είπα στις εναρτήριες παρατηρήσεις μου, προσπαθούμε να σεβαστούμε τις φορολογικές αρχές που έχουν αποφασιστεί από το Δικητικό Συμβούλιο και είμαι υποχρεωμένος να σεβαστώ. Κάθε φορολογικό μέτρο θα πρέπει να ληφθεί στα πλαίσια μιας κάποιας εμπορικής δραστηριότητας ανάλογα με τις εθιμικές εισαγωγικά πρακτικές οι οποίες ακολουθούνται στις διάφορες χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμε. Αυτό έχει σημασία νομίζω. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε εμείς το θέμα της, του προγραμματισμού στον τομέα της φορολογικής δραστηριότητας και η ευθύνη αναλαμβάνεται πάντα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το τμήμα που ασχολείται με φορολογικά δίδει συμβουλές σε όλες τις θεατρικές με βάση τον σεβασμό των αρχών που έχουμε δημοσιεύσει. Και έχουμε και την ευθύνη ακριβώς για τη λήψη των αποφάσεων αυτών. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα σε μια δεύτερη σειρά παρεμβάσεων από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Ντεμάζη από την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Δύο λεπτά. Ένα τραγούδι λέει Don't look back in anger, δηλαδή μη στρέφεις τα βλέμματά στο παρελθόν με οργή. Γι' αυτό και δεν θα πω τίποτα για το παρελθόν. Σας υπενθυμίζω όμως ότι καλείστε να πείτε την αλήθεια εδώ. Τα Χριστούγεννα να πάτε να πείτε στα παιδιά σα ό,τι θέλετε για του Άγιο Βασίλειδε. Και εγώ το κάνω άλλωστε. Εδώ όμω είστε υποχρωμένε και υποχρωμένοι να πείτε την αλήθεια. Ρωτώ λοιπόν, έρευνα τη Αμερικανική Γερουσία δείχνει ότι ένα κατασκευαστή. Ε, παιχνιδιών πλήρωσε 15 εκατομμύρια για φορολογική έρευνα για να μειώσει τα κέρδη του. Θα σας ρωτήσω όλες και όλους και αν δεν απαντήσετε σημαίνει ότι καταφάσκετε αν έχετε πληρώσει κάποιο τρίτο μέρος αν έχετε πληρώσει χρήματα σε κάποιον τρίτο μπορεί να είναι κάποια από τους Big Four, μεγάλους τέσσερις, ή και η φορολογική διοίκηση του, του Λουξεμβούργου ή κάποιες άλλες χώρες μέλους, αν έχετε πληρώσει λοιπόν κάποιον τρίτο. Αν δεν απαντήσετε, θεωρώ ότι απαντάτε καταφατικά. Δεύτερο, σας επισημαίνω την Amazon ιδίω ότι έχω γράψει γράμμα στον Bob Conford, ε, πρόεδρο του Tax, που είπε ότι το Λουξεμβούργο ήταν μέγας επιχειρηματικός εταίρος και ότι το Λουξεμβούργο και μάλιστα ο ίδιος ο πρόεδρος Γιούνκερ ως Πρωθυπουργό τότε του είχε προτείνει να του λύσει προβλήματα. Είστε διατεθειμένοι λοιπόν να απαντήσετε στο γράμμα αυτό και στο ερωτηματολόγιο του Bob Κόνφορντ, ο οποίος τώρα είναι επίτιμος πρόξενος του Λουξεμβούργου στο Σιάτλ. Τέλος, έχω μια ερώτηση για την HSBC το country by country reporting είναι ελληματικό. Πόσες θηγατρικές έχετε σε όλο τον κόσμο, πόσες από αυτές είναι απλές εταιρείες χρηματοκιβωτιού χωρίς καμιά σχέση με την οικονομική ζωή της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένες. Σας ευχαριστώ. Σβέν Γκίγκολτ από την ομάδα των Πράσινων. Ακούσαμε σήμερα ότι HSBC και Barclays είναι σύμφωνες με τη δημόσια country by country reporting. Θα ήθελα τώρα να ακούσω από Google, Amazon και Facebook αν μπορούν να αναλάβουν τη δέσμευση σήμερα στο μέλλον να δημοσιεύουν τα φορολογικά δεδομένα όπως και οι δυο που μόλις προανέφερα. Δεύτερο, είναι σημαντικό όντως εδώ στην Επιτροπή Τάξη να λέγεται η αλήθεια. Τα όσα είπατε για Google και Facebook για την χρήση των εταιριών σας στις Βερμούδες ή στα νησιά Καϊμάν είναι εξαπάτηση της Επιτροπής. Ασφαλώς και έχει επιπτώσεις στους φόρους που πληρώνονται στην Ευρώπη όταν με τη μεταφορά των κερδών φροντίζεται ώστε να μην γίνεται παραπέρα επιβολή φόρων στις πολιτείες Και μόνο με τη χρήση αυτών των θηγατρικών εταιριών μπορείτε να κάνετε φορολογικό dumping εδώ στην Ευρώπη. Τι έχετε να απαντήσετε. Δεύτερο, θα ήθελα να ακούσω ειδικότερα από την Google γιατί απέναντι στην SCC λέτε ότι έχετε μια σχετική εταιρεία στις Βερμούδες, στην ιστοσελίδα σας αναφέρετε 70 θηγατρικές, αλλά όχι αυτήν την, ε, ε, των Βερμούδων. Και από την HSPC πώς είναι τόσο μεγάλο ποσοστό το, φορο... το, το ποσοστό του κερδών σα στο Hong Kong που είναι γνωστός φορολογικός παράδεισος και περίπου από τα υπόλοιπα το 50% των κερδών σας από retail banking και wealth management είναι, ανακοινώνεται στο Hong Kong. Επίσης και τέλος για το Facebook. Εκτός από θηγατρικές σε Λουξεμβούργο, κάτω χώρες και Ελβετία. Μάλλον έχετε τέτοιες και αν ναι, γιατί. Μάρκο e Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ αναγνωρίζω την επιθυμία των εκπροσώπων των πιστοτικών ιδρυμάτων που είναι εδώ σήμερα να δεχθούν τις εκθέσεις αναχώρα, το country by country. Θα ήταν μια καλή κίνηση και ελπίζω αυτό να καταστήσει τη διαδικασία λεπτομερή και αποτελεσματική τα επόμενα χρόνια. Τώρα για τον εκπρόσωπο την HSBC εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο από το 2008-2009 γιατί βοήθησε πελάτες να δημιουργήσουν τρόπους ε, φορολογίας ιδιαίτερως ευνοϊκούς για αυτούς. Θα ήθελα, έχει περάσει λίγος καιρός από τότε και αναρωτιέμαι τι έχετε κάνει μέχρι τώρα έτσι ώστε αυτού του είδους τις συμπεριφορές να τις αποφύγετε. Πάντα σχετικά με τις τράπεζες. Θα ήθελα να καταλάβω γιατί είναι βολικό για αυτούς που εμπλέκονται στα χρηματοπιστωτικά να ελέγχουν ε, τα ταμεία τους ας πούμε σε περιοχές όπως το Λουξεμβούργο ή η Ιρλανδία και όχι σε άλλες χώρες. Ε, γιατί αυτό είναι πιο ευνοϊκό. Τώρα για τα Google, Facebook και Amazon. Θα ήθελα να μου διευκρινίσουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο αυτό που κάναμε στον προηγούμενο γύρο. Ε, τα stock options, πώς αυτό χρησιμοποιείται για να μειώνεται το φορολογικό εισόδημα. Ε, είπατε ότι εσείς αυτό είναι ένα πρότυπο ε, μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείτε για να, για να δίδετε αμοιβέ στους εργαζομένους εσάς. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφαιρείται ας πούμε από το ε, ενεργό κεφάλαιο της επιχείρησής σας και μειώνεται έτσι τον φόρο τον οποίο καλείστε να πληρώσετε πληρώνοντας υψηλές αμοιβέ. Και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαφορετικός τρόπος φορολογίας των κερδών σας και όχι γενικά με τον τρόπο με τον οποίο το κάνετε μέχρι τώρα. Ο κύριος Μονό, ο επόμενος ομιλητής. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν πρέπει να σας ευχαριστήσω εδώ για την παρουσία σας γιατί ακριβώς ε, σας απειλήσαμε για να έρθετε. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να μας υποτιμάτε. Μιας και ζούμε τις τελευταίες στιγμές αυτής της Επιτροπής, αποφασίσατε να θέσετε ένα τέλος σε αυτό το παιχνίδι του σκύλου και της γάτας. Εσείς θέλετε να συνεχίσετε το μόνιμο λόμπι σας και υποτίθεται ότι ξαφνικά είστε πρόθυμοι να συνεργαστείτε. Νομίζω λοιπόν ότι δεν είχατε ηθικά προβλήματα στο παρελθόν όπως και τα Starbucks και η Fiat και η HSBC ε, χρησιμοποίησατε πολλές μεθόδους για το πλήσιμο ε, χρημάτων και στην Ελβετία ακόμα και μεξικανικά χρήματα ε, έσοδα από ναρκωτικά, από εμπόριο ναρκωτικών η Barclays δεν έχει μείνει πίσω από αυτού τους δραστηριότητες, αν και δεν έχει δραστηριοποιηθεί τόσο πολύ. Πράγματι η Amazon αυτή τη στιγμή καθυστερεί τις πληρωμές της στην Γαλλία, γιατί υποτίθεται ότι βρίσκεται υπό έρευνα στο Λουξεμβούργο. Νομίζω ότι έτσι θα συνεχίσετε να δημοσιεύετε τα προσωπικά στοιχεία των πολιτών σας χωρίς προειδοποίηση. Βασικός στόχος φυσικά είναι η χρηματοδοτική αποδοτικότητα. Δεν έχει σημασία το συμφέρον των πελατών σας, αλλά θέλετε απλά να προστατεύσετε τα συμφέροντα των δισεκατομμυριούχων. Το οικονομικό ε, παγκοσμιοποιητικό αν θέλετε καπιταλιστικό σύστημα σας το επιτρέπει. Ε, αν ξαφνικά περάσουμε τώρα σε μια νέα κατάσταση όπου θα, παρουσιαστούτε με, θα παρουσιαστείτε με κατάλληλες συνειδήσεις, τότε ε, νομίζω ότι πάλι τα κράτη και οι πολίτες δεν θα πρέπει να σας πιστέψουν. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε και πάλι όπως και πριν με την Google. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ε, αρχίσω με την πρώτη ερώτηση με την εμπλοκή τρίτου μέρους. Αν δείτε την φορολογική δομή και πώς ε, σε μια πολυεθνική εταιρεία ε, είναι δομημένο το τμήμα που ασχολείται με τις φορολογικές υποθέσεις φυσικά υπάρχει τρόπος ελέγχου θέλουμε να ξέρουμε τι λειτουργεί καλά και τι δεν λειτουργεί και φυσικά φροντίζουμε να συμμορφωθούμε με την νομοθεσία όλων των κρατών στα οποία ε, δραστηριοποιούμαστε και δεν νομίζω ότι είναι προβληματικό να χρησιμοποιούμε σύμβουλες ε, τρίτων. Ο κύριος Θεμαζή, μα δεν ρώτησα αυτό, εγώ ρώτησα εάν έχουν υπάρξει αμοιβέ που ε, είναι αναλογικές με τους φόρους στους οποίους γλιτώσατε χάρη σε αυτές τις ε, συμβουλές. Επαναλαμβάνω, λέει ε, απαντώντας ο μιλητής, ότι δεχόμαστε συμβουλές ε, ούτως ώστε να συμμορφωθούμε με την ομοθεσία των χωρών όπου δραστηριοποιούμαστε. Άρα συνάγω ότι συμφωνείτε με τη διαπίστωσή μου, λέει ο κύριος Τεμάζη. Καμία απάντηση. Τώρα θα ήθελα, λέει ο να ε, σχολιάσω το θέμα των εκθέσεων αναχώρα. Όλοι είμαστε υπέρ της διαφάνειας ε, και σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δημοσιεύουμε τους φόρους που καταβάλουμε θα πρέπει να δείτε ότι υπάρχει και η συμφωνία μεταβίβασης ε, της φορολόγησης ε, σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία ε, που διέπει τη σχέση μητρικής με θηγατρικές. Ε, ε, υπάρχουν λοιπόν ε, εταιρείε συμβουλών σε χώρες και αυτό αναφέρεται κάθε φορά στη δημοσίευση των πληροφοριών. Βλέπουμε όμως και πάλι, και το τονίζω γιατί είναι βασική αρχή, ότι καταβάλουμε τους φόρους σε σχέση με τα κέρδη μας και όχι σε σχέση με το εισόδημα. Η διαφάνεια στο φορολογικό σύστημα ε, σίγουρα είναι μια αρχή που ανστερνιζόμαστε όλοι. Διακόπτει ο κύριος ε, Κίκολτ. Εσείς αναλαμβάνετε τη δέσμευση να υποβάλλετε εκθέσεις αναχώρα. Απάντηση βάσει των ε, κανόνων και βάσει της ε, συμφωνίας μετατόπισης της φορολόγησης arm's length υποβάλλουμε εκθέσεις. Αυτό δεν είναι καμία απάντηση λέει ο κύριος Κίκολτ. Δεν υποβάλλετε τέτοιες εκθέσεις όπως στις τράπεζες. Απάντηση. Μα εξαρτάται από την νομοθεσία των κρατών. Σε κάποιες χώρες είναι δημόσιες αυτές οι πληροφορίες. Μπορείτε εσείς όμως να αναλάβετε, λέει ο κύριο Γκίγκολ, δέσμευση, γιατί εσείς αποφασίζετε πώς υποβάλλετε τις εκθέσεις. Εμείς αναλαμβάνουμε, απαντάει ο πρόσωπος του Google, ε, να ε, τηρούμε την νομοθεσία των κρατών μελών και βάλουν οι κυβερνήσεις. Ε, πρόεδρος, Σα έχει απαντήσει, κύριε Γκίγκολ, ή δεν είναι η απάντηση που θέλετε, αλλά ε, έχει δοθεί μια απάντηση από τον εκπρόσωπο της Google. Και φυσικά θα συμμορφωθείτε με την νομοθεσία. Τέταρτη ε, απάντηση, ε, και αυτό σχετίζεται και με την ερώτηση του κύριου, ε, χρειαζόμαστε κανόνες για να υπάρχει συμμόρφωση. Νομίζω ότι αυτά τα ε, ηθικά ζητήματα θα πρέπει να τα τακτοποιούμε μέσω της νομοθεσίας ε, και οι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν ε, να είναι οι ίδιοι για όλους, για τις πολυεθνικές και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστούμε κυρία Διακόπτω πάλι ο κύριος Γκίγκλ. Για την Σβερμούδα σας έκανα και μια άλλη ερώτηση και δεν απαντήσατε. Μπορείτε να την επαναλάβετε. Ναι, έλεγα ότι κατα... υποβάλατε ψευδή δήλωση λέγοντας ότι η δομή στις Βερμουδές ε, δεν έχει καμία σχέση με την εφορολογική σας ε, αποφυγή. Ε, δεν ισχύει αυτό διότι εάν ίσχυαν οι αμερικανικοί φορολογικοί συντελεστές ε, θα είχατε απολέσει κάθε κέρδο. και άρα δεν ευσταθεί αυτό που είπατε. Απάντηση. Ε, στην ε, Βερμούδα είπαμε ότι έχουμε αναβολή ρύθμιση των φορολογικών υποχρεώσεων και άρα η βάση αυτής της συμφωνίας μετατόπισης της φορολόγηση σε arm's length αυτό κάνουμε ακριβώς, δηλαδή κρατάμε τα χρήματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα επενδύουμε στην Ευρώπη, δισεκατομμύρια επενδύουμε στην υποδομή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ε, γίνεται χάρη στο ότι δεν ε, έχουν αναβληθεί οι φόροι στις ΕΠΑ. Ναι, αλλά έπρεπε να καταβάλλεται υψηλότερο εταιρικό φορολογικό συντελεστή στις ΕΠΑ. Ε, έτσι φοροδιαφεύγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο διότι κάνετε την αναβολή ε, της ρύθμισης των φορολογικών ε, υποχρεώσεων μέσω της θηγατρική τη Βερμούδης. Να είστε ειλικρινεί. Απάντηση. Σας είπα ότι ε, εφαρμόζεται αυτό το μοντέλο μετατόπιση ε, ε της, της σε arm's length και ε, θα έπρεπε να διορθωθεί αυτό, αλλά αυτό θα το αποφασίσουν οι κυβερνήσεις βάσει των κανόνων του ΩΣΑ. Προς το παρόν ισχύει αυτό το μοντέλο, Πρόεδρος. Γι' αυτό το λόγο σας ερώτησα προηγουμένως αν θα μπορούσατε να είστε συγκεκριμένοι και να μας υποβάλλετε γραπτός τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας σε σχέση με τις, τον αντίκτυπο ε, αυτών των συμφωνιών ε, για τους φορολογουμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός και στις ΥΠΑ αφετέρου. Ε, μπορείτε να απαντήσετε και στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Νομίζω ότι ολοκλήρωσα. Ε, κύριε Ρον, ε, ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα. Για τα third parties, συμβουλές από τρίτα μέρη. Ναι, χρησιμοποιούμε συμβούλους για τους ίδιους λόγους που εξέθεσε και ο εκπρόσωπος της Google. ούτω ώστε να συμμορφωνόμαστε πλήρω με την νομοθεσία κάθε χώρα Έχουμε ε, μία ομάδα για τα φορολογικά ζητήματα στην εταιρική μας ε, έδρα που δεν γνωρίζει όμως απαραίτητα τους φορολογικούς κανόνες στην επικράτεια όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ως εκ τούτου καταφεύγουμε σε συμβουλές τρίτων. Το θεωρούμε φυσιολογικό. Σε σχέση τώρα με την υποβολή εκθέσεων αναχώρα, διακόπτει ο κ. Δεμασκή πάλι, δεν ήταν αυτό που σας ρώτησα. Εγώ σας ρώτησα εάν αν αμείβεται τα τρίτα μέρη σε ε, σχέση αναλογικά με, τα, με τους φόρους που γλιτώσατε χάρη στη συμβουλή σας. Ο γιος μου είναι εξάχνος και θα μπορούσε να καταλάβει αυτό το ερώτημα. Εσείς δεν μπορείτε. Απάντηση. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Αν καταλαβαίνω καλά, μας ρωτάτε εάν αν αμείβουμε τους συμβούλους βάσει της αποτελεσματικότητάς τους ε, ως προς την εξοικονόμηση φορολογική. Ε, μπορείτε να μας απαντήσετε γραπτός, λέει ο πρόεδρος, βεβαίως, ένα πρόβλημα. Γιατί είναι υποβολή εκθέσεων χώρα Δυστυχώς θα είμαι νεαρή και θα επαναλάβω αυτά που σας έλεγα προηγουμένως. Συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις διαφάνειας που ισχύουν ε, στις διάφορες χώρες. Δημοσιεύουμε τις απαιτούμενες ε, βάσει της κείμενης νομοθεσίας ε, πληροφορίες. Εάν ένα μοντέλο υποβολή εκθέσεων αναχώρα ισχύσει για ολόκληρη την Ευρώπη, φυσικά και θα συμμορφωθούμε με αυτού τους κανόνες. Για το θέμα των ε, νήσων Καϊμάν, μιλήσατε για φορολογικό ντάμπινγκ. Και πάλι θα διαφωνήσουμε ε, με αυτήν την... Ε, περιγραφή της κατάστασης, ε, διότι πρόκειται για αναβολή ρύθμισης ε, φορολογικών υποχρεώσεων ως προς τη ΣΥΠΑ και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζονται χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με εξαίρεση την Ιρλανδία και ως προς την Ιρλανδία συμμορφωνόμαστε πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία και το ίδιο θα κάνουμε και στο μέλλον όταν, θα όταν θα να ισχύει τροποποιημένη νομοθεσία. Για τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, στην Ολλανδία έχουμε ε, υποκατάστημα, στην Ελβετία όχι, ε, στο Λουξεμβούργο έχουμε μια νομική οντότητα και αυτά ε, και αυτό είναι όλο. Επειδή τώρα δεν μπορώ να σας κοιτάω κιόλας για να σας απαντήσω, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Δυσκολεύομαι με το μικρόφωνο. Αυτά τα stock options είναι ένας τρόπος αμοιβή και, για τις, και στις startup εταιρείε χρησιμοποιείται. Είναι πολύ ελκυστικό ακόμη και για τις πολύ καινοτόμες ε, νέες εταιρείες που δεν έχουν απαραίτητα τα μέσα ε, να ε, προσελκύσουν ε, προσωπικό με τις αμοιβέ και άρα τους προσελκύουν ε, καθιστώντας τους μέτοχους. Στη Γαλλία, στη χώρα μου, θεωρείται αυτό ένας ε, παράγοντας καινοτομίας για την οικονομία. Είναι ένας παράγοντας έλξης και είναι σημαντικό για την οικονομία. Σας ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μακίνων. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, κάθε φορά σας ξεχνώ. Ο κύριος Ντίσμεν. I'm sorry. I'm sorry. Um, coming back to the country by country. Για την έκθεση αναχώρα και τις ερωτήσεις που τέθηκαν, όπως είπαμε, υποστηρίζουμε την μέθοδο αυτή είναι βασικό μέσο εκτίμησης αξιολόγησης κινδύνου. Έτσι ε, θα κατανοήσουμε όλοι καλύτερα τα φορολογικά θέματα των επιχειρήσεων ανά χώρα. για το αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημοσιοποιείται. Δεν νομίζουμε, για διάφορους λόγους. Καταρχάς, αν δεν υπάρξει επιπλέον επεξηγηματικό περιεχόμενο, η πληροφορία μπορεί να είναι παραπλανητική στην αναγνωσή της. Δεύτερον, συνήθως τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν εμπιστευτικά στοιχεία επιχειρηματικά, κέρδη κτλ. Δεν είμαστε υπέρ της δημοσιοποίησης των εκθέσεων αυτών. Για τους tax consultants φυσικά και έχουμε χρησιμοποιήσει σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε εμπειρογνώμονες δικούς μας, υπαλλήλους δικούς μας σε όλες τις χώρες που να ελέγχουν το νομικό πλαίσιο, το μελλοντικό ή το ισχύον. Τους πληρώνουμε να κατανοήσουν, όχι να βρούνε τους ευνοϊκότερους όρους. Ένα απλό παράδειγμα, όταν πηγαίνει κάποιος σε μια νέα χώρα πρέπει να πάρει μια απόφαση αν θα πρέπει να χρηματοδοτήσει κάτι με ε, συγκεκριμένα κεφάλαια ή με αποδείξεις χρέους. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έχει διαφορετικές συνέπειες σε φορολογικό επίπεδο. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κάποιος να μας συμβουλεύσει. Ε, εγώ δεν έχω δει μια κατάσταση στην Amazon όπου να ισχύει κάτι ε, τέτοιο που, είπε, που ανέφερε ο κύριος βουλευτής. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό. Η τρίτη ερώτηση αφορά τις αποζημιώσεις ή αντισταθμίσεις αν θέλετε. Ε, υποτίθεται ότι χρησιμοποιούμε το μέσο αυτό για να μειώνουμε το φόρο. Όχι, η πληρωμή με μερίσματα, με μετοχές είναι βασικό ε, τμήμα της δραστηριότητας των μεγάλων επιχειρήσεων εμείς έχουμε πάρα πολύ στην Amazon, αυτοί που εργαζόμαστε, την αίσθηση της ιδιοκτησίας στην επιχείρηση και γι' αυτό μας πληρώνουν και με α, μετοχές. Ο, ο εκπρόσωπος των τραπεζών τώρα, κ. Μακίνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πέντε ερωτήσεις μου έχουν τεθεί, στις οποίες θα σταθώ σύντομα. Η πρώτη ερώτηση για το αν χρησιμοποιούμε συμβούλους και αν πληρώνονται σε σχέση με τα κέρδη τα οποία μας επιτρέπουν να έχουμε. Όχι. Υπάρχουν τομείς στους οποίους ο σύμβουλος δεν δίνει τις υποχρεωτικά καλύτερες σύμβολες, οπότε θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε και δεν θεωρούμε ότι κάθε τι το οποίο λέγεται από πλευρά συμβούλων είναι δεδομένο. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να δεχτούμε, εγώ προσωπικά, όπως επίσης και οι υπόλοιποι υπεύθυνοι για τα φορολογικά, τέτοιου είδους α, ιδέες δεν τους ικανοποιούν. Δεύτερο, πόσες θηγατρικές έχουμε και πόσες από αυτές είναι απλά γραμματοκιβώτια. Ο αριθμός των θηγατρικών που έχουμε θα τις δημοσιεύσουμε στο τέλος του χρόνου επίσημα. Είναι περίπου 800 σε παγκόσμιο επίπεδο, ήταν 1500 πριν 6 χρόνια και στόχος μας είναι να μειωθεί ο αριθμός αυτός σε 600 ίσως 550 μέχρι το τέλος του 16 2017 ίσως. Ε, ε, ε, επιχειρήσεις γραμματοκιβώτιο. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείται με αυτό. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις θηγατρικές για να διοχετεύουμε τα κέρδη από εκεί όπου τα βγάζουμε. Ο στόχος των θηγατρικών είναι ακριβώς να καλύπτουν τις ειδικέ καταστάσεις στην περιοχή τους όταν υπάρχουν, αλλιώς καταργούνται και με τις διαδικασίες ελέγχου ε, ξεπλήματος ε, του ε, βρώμικου χρήματος κανένας δεν έχει συμφέρον να κρύβεται. Η διαφάνεια η φορολογική είναι βασικός μας στόχος και το να πληρώνουμε δίκαια επίπεδα φορολογίας στις χώρες όπου δραστηριοποιούμεθα είναι σωστό. Είναι μια τεράστια επιχείρηση η HSBC, η αρχική της έδρα ήταν στο Hong Kong Ήρθαμε στην Ευρώπη ε, τα τελευταία 20 χρόνια μόνον. Ε, δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο για μας ε, το να δραστηριοποιούμεθα σε αυτό που ονομάζουμε εξωτικές χώρες, αλλά έχουμε πραγματικές εργασίες, έχουμε πραγματικό τζίρο σε εισαγωγικά σε αυτές τις χώρες και εκεί προσπαθούμε να πληρώσουμε το φόρο ο οποίος μας αναλογεί με δικαιοσύνη και δεν χρησιμοποιούμε ψευδεπίγραφες επιχειρήσεις. Έχετε υπαλλήλου σε όλες τις χώρες, σε κάθε μία από αυτές τις θηγατρικές βεβαίως. Και φυσικά μπορούμε να σας δώσουμε ε, τις εκθέσεις αναχώρα για το 2014 και μπορώ και αμέσως μετά την συνεδρίαση να σας δώσω τα στοιχεία. Ε, τώρα για λόγους χρόνου. Ε, αυτά που είπε για τα κέρδη και το Χονγκ Κόνγκ. Είπαμε ότι αυτή ήταν η αρχική μας έδρα. Δημιουργηθήκαμε εκεί μετά το Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο. Ήμασταν η μεγαλύτερη τράπεζα εκεί, σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την περιοχή. Είμαστε υπερήφανοι. Όταν πάτε στο Χονγκ Κόνγκ θα δείτε την έδρα μας, το κεντρικό μας κτίριο. Ε, χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται εκεί και χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται γενικά στην Άπο Ανατολή τι είναι η βασική μας δραστηριότητα και είμαστε υπερήφανοι για αυτήν. Η επόμενη ερώτηση, τι διαφορά ε, υπάρχει στο λεγόμενο private banking. Αν έχουμε αλλάξει τις αντιλήψεις, πράγματι έχουμε μειώσει τον αριθμό των πελατών σε αριθμούς που μπορούμε να διαχειριστούμε με ασφάλεια. Προσπαθούμε επίσης να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το private banking λειτουργεί με πλήρη φορολογική διαφάνεια. Τώρα, γιατί να χρησιμοποιήσουμε το Λουξεμβούργο. Αυτό το συζήτησα και με τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε έδρες ταμείων και ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά υπάρχουν θέματα και διοικητικά και φορολογικά τα οποία μας εμποδίζουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε με την αρμόδια ελεγκτική αρχή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περνάμε στον τελευταίο γύρο των ερωτήσεων. Δίνω το λόγο στον κύριο Νίντε Μάγερ για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δύο λεπτά. Διακόπτει ο πρόεδρος. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ξέχασα την τράπεζα Barclays, κύριε Χεράρτ. Δύο ερωτήσεις μου έκαναν τα μέλη σας απάντησε σε ίδια ερώτηση και ο κύριος ε, Μακίναν για το Λουξεμβούργο και για τα φαντς ε, εκεί. Είμαστε χρόνια στο Λουξεμβούργο, εμείς οι Barclays, γιατί είναι μέγα ε, κέντρο. Έχουμε και άλλες τράπεζες εκεί, έχουμε πελάτες εκεί, υποστηρίζουμε, υποστηρίζει το Λουξεμβούργο την, τον χρηματοπιστωτικό κλάδο Γι' αυτό ε, το, ε, την αναβολή φόρων, ε, τους αναβαλόμενους φόρους, δηλαδή αυτό δεν το αναγνωρίζω. Για το θέμα των συμβούλων. Χρησιμοποιούμε συμβούλους, τις υπηρεσίε συμβούλων δηλαδή, όπως εξήγησε και εκπρόσωπος της Amazon. Δεν έχω γνώση για αμοιβή τους αναλόγως με τα φορολογικά έσοδα που μας γλιτώνουν, τα φορολογικά ε, τους φόρους που μας δηλαδή. Όπως έχω ξαναπεί, προ δύο ή τριών ετών επιβάλαμε ένα σετ φορολογικών προτύπων που το 2013 δηλαδή, που τα, τα επιβάλλουμε σε όλες τις τραπεζές μας. Αυτό νομίζω ότι σας απαντά. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Τότε, τελευταία σειρά ερωτήσεων Τώρα είστε σίγουρος κύριε Πρόεδρε ότι είμαι εγώ. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήλθατε. Από την Amazon είπε η εκπρόσωπος ότι η σαφήνεια είναι πολύ σημαντική και ο επικεφαλής του φορολογικού τμήματος της Barclays μίλησε για το σχέδιο BEPS και για το CCCTB του ΟΣΑ δηλαδή και της Επιτροπής. Εγώ συμφωνώ με την άποψη ότι η σαφήνεια είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως και η σε εφαρμογή των κανόνων. Δύο ερωτήσεις. Πρώτη, ποιο τμήμα του σχεδίου του ΟΣΑ για το BEPC σας φαίνεται το πιο σημαντικό για την αύξηση της διαφάνειας για την εφαρμογή των φορολογικών κανόνων και ποιο τμήμα σας ανησυχεί. Δεύτερο, έλλειψη διαφάνειας δεν ε, χαρακτηρίζει μόνο τους εθνικούς φορολογικούς κώδικες, καμιά φορά προκύπτει και από τις διαφορές και μεταξύ των εθνικών φορολογικών κωδίκων. Νομίζω ότι η πρόταση της κοινή ενοποιημένη φορολογικής βάσης για τις επιχειρήσεις που έγινε πριν από δύο χρόνια νομίζω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σημαντικό βήμα και το έχει υποστηρίξει και το Ευρωκοινοβούλιο για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Ποια είναι η άποψή σας και συνιστάτε στις κυβερνήσεις να το στηρίξουν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Λουντεκ. Η κυρία Φερέιρα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η οποία μάλιστα είναι και συνεισηγήτρια και αυτή. Μάλιστα, να σας τα πω στα αγγλικά για να με καταλάβετε πιο εύκολα. Για το Google πρώτα. Είπατε ότι δηλώνεται Όμως 8,8 δισεκατομμύρια μεταφέρατε στις Βερμούδες σε ένα νησί δηλαδή που έχει 16.000 κατοίκους. Δεν ταιριάζει με την φορολογική σας δήλωση και αναμένουμε την απάντησή σας σχετικώς με, τον, με ποια φορολογική αρχή ε, προσπαθείτε να φοροαποφύγετε την Αμερικανική ή την Ευρωπαϊκή. Σε ό,τι αφορά τώρα εσάς Facebook εξεπλάγει από την πληροφορία που δώσατε ότι ενισχύσατε πολλές πληρωμές στο Ενωμένο Βασίλειο διότι κατά μέσον όρο για το 2014 ε, δίνεται 210.000 λίρες τερλίνες ανά έτος, αυτός είναι ο μέσος όρος δηλαδή των ε, αμοιβών που δίνεται και πληρώσατε φόρο 4.037 λίρες τερλίνες. 4.000 λίρες. Άρα δηλαδή δεν καταβάλλετε φόρους εκεί όπου δημιουργείται αξία. Αφού λοιπόν δεν δημιουργείται αξία από τις, από τις δραστηριότητες σας στο Ηνωμένο Βασίλειο, τότε γιατί έχετε εκεί οτιδήποτε, οποιαδήποτε λειτουργία. Και γιατί έχετε μια αντιτέ μια νομική οντότητα, δηλαδή στο Λουξεμβούργο είναι και ενώ έχετε απλώς ένα γραφείο στις βαλτικές χώρες. Αυτά είπατε ποιος είναι ο ρόλος αυτών των οντοτήτων, διότι αν δεν δημιουργείται πλούτος εκεί, αν δημιουργείται αξία δηλαδή, τότε ποιος είναι ο λόγος. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι κινήσεις. Για την Barclays τώρα. Θα ήθελα να γνωρίζω πόσες ακριβώς δραστηριότητες έχετε στις ανεξάρτητες νήσους. Σας ευχαριστώ. Λαϊκό κόμμα, κύριος Κίρτσος. President. Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις. Το φορολογικό σύστημα για τις εταιρείες σας ε, στις Είπα, είναι λιγότερο ή περισσότερο αυστηρό σε σχέση με αυτά ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. μπορείτε να κάνετε μια σύντομη σύγκριση ανάμεσα στα δύο για τη φορολόγηση των κερδών πρώτων και δεύτερον για να προωθήσετε τη μακροπρόθεσμη φορολογική στρατηγική των εταιριών σας. Ε, προσπαθείτε να αποδείξετε ότι είστε φιλικοί προς τους ε, πελάτες. Το ίδιο ισχυρίζεστε και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες σας και θέλετε να λάβετε δέσμευση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη για να, να έχετε μια μεγαλύτερη συμβολή για την καταπολέμηση της στόχης και των κλιματικών αλλαγών στις ε, χώρες όπου επικεντρώνονται οι δραστηριότητες ε, και τα κέρδη σας, ε, γιατί δεν μπορείτε να είστε φιλικοί με τους καταναλωτές σας, κοστίζει πολύ ή θεωρείτε ότι δεν ασχολούνται οι άνθρωποι με το ποιος πληρώνει φόρους που δεν θα θέλατε οι εταιρείε σας να είναι φιλικότερες προς τους Ευρωπαίους φορολογουμένους ή μήπως αυτό δεν είναι μέρος της φορολογικής σας στρατηγικής. Σας ευχαριστούμε. Και η Ευελίν Ρέγνερ τώρα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ε, να απευθύνω το ερώτημά μου στον κύριο Χαβέρτ προς την Βάρκλε. Ε, πόσες ε, έχετε σε υπερπόντια εδάφη και ε, ε, εδάφη της κοινοπολιτείας προς την Facebook. Προσπαθούμε να, με διάφορους τρόπους να ε, έχουμε πιο ξεκάθαρες ε, ε, πληροφορίες από πλευρά σας. Όταν μιλάτε για τον ουσιαστικό φορολογικό συντελεστή λέτε ότι αφορά το 40% των κερδών σας. Τι εννοείται ακριβώς με αυτό το 40% και τώρα για την υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Πόσα ε, επενδύεται για λόμπινγκ σε άτομα, σε προσωπικό, σε λεφτά ε, για τους ηθήνοντες, ε, για τους πολιτικούς και για όσους ασχολούνται με την υποβολή εκθέσεων ή φορολογικά ζητήματα. Για την διαβούλευση για το BEPS λάβαμε πάρα πολλές ε, απαντήσεις ε, από εταιρείες. Ε, με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι δραστηριότητες lobbying που έχει η Facebook σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να αλλάξουμε την σειρά με την οποία θα απαντήσουν οι ομιλητές για να έχουμε μια καλύτερη ισορροπία. Ο κύριος Κερμπέν και έτσι δεν θα τον ξεχάσω κιόλας όπως το περασμένο γύρο. Έχετε ερωτήσεις συγκεκριμένα για την Barclays. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα αρχίσω με αυτές τις ε, δύο τελευταίες ερωτήσεις ε, ε, στα, για την παρουσία μας στα υπερπότια εδάφη και σε χώρες κοινοπολιτείες. Οι δραστηριότητες μας και τα ποσοστά φαίνονται στη, στα στιγμιότυπα στις εκθέσεις αναχώρα για κάθε μία από αυτές τις χώρες όπου προσφέρουμε διάφορες ε, υπηρεσίες επενδυτικές, μεσητείας, ε, λιανικής, τραπεζικής και το καθεξής. Ε, ο αριθμός των θηγατρικών μας 14 στο Γκέρσι, στο ΕΛΟΦΜΑΝ 23, στο Γκέρσι 24. Απασχολούμε πάρα πολλούς ανθρώπους και σε αυτά τα δύο νησιά. Ήθελα επίσης σε σχέση με τον Όμιλο να μου πείτε ακριβώς πώς, τι ποσοστό κερδών δηλώνεται εκεί. Για το 2014, για τα κέρδη 2.34 για το Jersey και 117 στην είσοδο του Μαν Και αυτά είναι τα ομαδοποιημένα στοιχεία. Οτιδήποτε είναι κάτω αυτού δεν αναφέρεται. Ε, σας είπα ότι βλέπετε το στιγμιότυπο στην έκθεση αναχώρα. Ε, βλέπετε ακριβώς τον αριθμό των εργαζομένων σε κάθε θηγατρική ε, σε αυτή την έκθεση. Για το πρώτο ερώτημα, για το BEPS και την ε, κοινή βάση φορολόγησης. Νομίζω ότι η πιο χρήσιμη πτυχή του BEPS είναι ότι θα έχουμε μεγαλύτερη συνέπεια, λιγότερες διαφορές, ισότιμους όρους ανταγωνισμού ε, και νομίζω ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση με τον τόπο φορολόγησης ε, των κερδών ε, και ούτως ή άλλως αυτή την προσέγγιση έχουμε υιοθετήσει και στην Barclays. Αυτό το σύστημα της, ε, των εκθέσεων αναχώρα το έχουμε προωθήσει ούτως ή άλλως περισσότερο και νομίζω ότι οι κυβερνήσεις θα μπορούν να αξιολογήσουν τους κινδύνους χάρη σε αυτές τις αυξημένες πληροφορίες. Ε, κατά πάσα πιθανότητα για ε, φόρους ε, για φορολόγηση των εισοδημάτων ε, και για ενδεχόμενες διαμάχες για διπλή φορολόγηση ή διαφορές ανάμεσα στις κυβερνήσεις και τις εταιρείες, κάτι που θα είναι φυσική απόρρια της ισχύω του νέου συστήματος, θα χρειαζόμασταν και ένα σύστημα διαιτησίας. Ξέρω ότι υπάρχει ομάδα των 20 που έχουν ήδη εκφράσει ε, την επιθυμία τους να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο σύστημα και φυσικά όσο περισσότεροι δηλώσουν θα το υποστηρίξουν τόσο καλύτερα. Για την κοινή ε, ε, την ενοποιημένη βάση φορολόγηση CCTB η κοινή βάση θα ήταν κάτι απλούστερο, δηλαδή θα είχαμε ε, ίδιους κανόνες σε 28 κράτη-μέλη. Αυτό θα είχε απλουστεύσει τη το σύστημα. Όμως, όπως αναγνωρίζει και η δική σας η Επιτροπή στην έκθεσή της, αυτό προϋποθέτει μεγαλύτερη εναρμόνιση των ε, ε, λογιστικών προτύπων ε, στα οποία βασίζεται αυτό το σύστημα. Νομίζω ότι ε, η μέτρηση των φορολογητέων κερδών βάσει αυτών των κοινών λογιστικών προτύπων είναι το βασικό πρόβλημα. Προτού καταλήξουμε στην ενοποιημένη βάση και φυσικά το, ε, το πώς διαχειρίζονται τη φορολογική πολιτική οι οι φορολογικές αρχές. Τώρα για την ενοποίηση του CCTB πέρα από την ε, κοινή βάση δηλαδή Νομίζω ότι οι επιχειρήσεις ε, θα ήταν υπέρ ενός τέτοιου συστήματος, όμως αυτή η συμφωνία του Arms Length για τη μετατόπιση της τιμολόγησης θα συνεχίσει να ισχύει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε προσοχή. Πώς ποιον αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό και νομίζω ότι τελικά αντί να πλουστεύσουμε μπορεί να περιπλέξουμε το σύστημα για ομίλους όπως η Barclays παραδείγματο χάρη που ε, δραστηριοποιείται σε πολλές περιοχές του κόσμου. Και άρα θα πρέπει να λειτουργεί βάσει διαφορετικών συστημάτων. πρόεδρο ευχαριστούμε. Όντως, ε, θα είναι πάρα πολύ περίπλοκο το ζήτημα και θα πρέπει να το ε, συζητήσουμε με τους ομοτήμους μας στον ΟΣΑ. Ο κύριος Μακίνων. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την CCCTB, την ενοποιημένη βάση. Θα ήθελα να ευεώσω αυτά που είπε ο συνάδελφος από την Barclays. Ζητούμε ενάργεια και διαφάνεια. Αν επιστρέψουν λοιπόν στις βασικέ αρχέ των λογιστικών προτύπων, στην έκθεση BEPS εξάλλου μιλάμε για την ε, συνοχή, την συνέπεια και τη διαφάνεια ως προς τα λογιστικά πρότυπα. Αν λοιπόν το CCCTB μας δώσει ε, περισσότερη διαφάνεια θα ήμασταν πρόθυμοι να το υποστηρίξουμε. Ε, τώρα σε σχέση με την υιοθέτηση ενό ευρωπαϊκού συστήματο, αν υπεκρατήσει η διαφάνεια, δεν, έχουμε, δεν μπορούμε να είμαστε εναντίον, εκτό και αν αυτό οδηγεί σε άδικη φορολόγηση ή διπλή φορολόγηση εάν ε, καταφέρνουν ε, οι κυβερνήσεις να καταλήξουν σε ένα εύρυθμα ε, σε ένα εύρυθμο σύστημα το οποίο θα εφαρμόζεται και σωστά, τότε δεν θα έχουμε καμία ένσταση. Για το BEPS νομίζω ήταν πολύ λογικά αυτό που μας είπε ο συνάδελφος. Οι τομείς που μας απασχολούν στην, στις χρηματοοικονομικές αγορές είναι ε, οι πληρωμές που γίνονται, διότι ε, ο δικός μας ο τομέας υπάγεται σε πολύ αυστηρές ρυθμίσεις Οπότε οποιοδήποτε περιορισμό θα πρέπει να είναι ε, διόντως αιτιολογημένος. Πρέπει όμως να λαμβάνεται υπόψη και η δομή του τραπεζικού τομέα. για, από τον ΩΣΑ για την εφαρμογή του BEPS. Επίσης, χρειαζόμαστε περισσότερα πολυμερή μέσα, διότι χάρη σε αυτά θα επικρατήσει ε, μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με το τι ζητούν ε, οι φορολογικές αρχές, όπως ε, υπάρχει το θέμα των φορολογικών διαφορών στην HSBC παραδείγματος χάρη προσπαθούμε να μεταφέρουμε μία πρακτική σε κάποια άλλη, ε, στην επικράτεια κάποιας άλλης χώρας και βλέπουμε ότι απαγορεύεται αυτό ε, λόγω ε, των έμεσων φόρων παραδείγματος χάρη για τις υπηρεσίες ή άλλα φορολογικά εμπόδια που συναντούμε και δεν μπορούμε να θεωρήσουμε δηλαδή ότι για τις υπηρεσίες ισχύει το ελεύθερο εμπόριο για μας αυτό είναι πηγή ανησυχίας. Ε, το BEPS δεν ρυθμίζει λοιπόν αυτό το ζήτημα και άρα χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό διευθέτησης των διαφορών. Ε, και δεν θα ήθελα τώρα να επεκταθώ. Ε, καλή τύχη εύχομαι, διότι είναι τρεις βασικές αρχές της, του BEPS και συμφωνούν με, την, με τον προσανατολισμό της HSBC. Πρόεδρος. Έχετε δίκιο να επιμένετε στο σύστημα επίλυσης διαφορών είναι ένα θέμα το οποίο τα ομόσπονδα κράτη, τα οποία έχουν επιχειρηματικό φόρο και σε επίπεδο κεντρικού κράτους και σε επίπεδο ομοσπονδιακών δομών, έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν Ελβετία, Καναδάς και Ηνωμένε Πολιτείε. Το Amazon ίσως δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι. Σας ευχαριστώ στα θέματα πολιτικής και σε ποιους τομείς τα ε, ε, θέλαμε να κρίνουμε ότι τα BEPS είναι σημαντικά. Η, φυσικά η κοινή επιχειρηματική η φορολογική βάση. Απαιτούνται εδώ να υπάρξουν ορισμένες διευκρινήσεις, απαιτείται προσπάθεια τους επόμενους ε, μήνες και για τον ΠΕΠΣ στον ΟΣΑ σε σχέση με την κατανομή των κερδών γιατί αν αυτό δεν είναι κάτι το θα έλεγα ξεκαθαρισμένο εμείς ως φορολογούμενοι βλέπουμε ότι μπορεί δυνητικά να υπάρξει κάποιος κίνδυνος. Υπάρχουν επίσης κάποιοι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών οι οποίοι πρέπει να είναι τοπικοί ή έστω περιφερικοί έχουν και αυτή μεγάλη σημασία. Υπάρχουν στοιχεία στο εσωτερικό των BEPS ε τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν για μας προτεραιότητες. Αν συγκρίνουμε το φορολογικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών με το ευρωπαϊκό, είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να συζητήσουμε σε τρία λεπτά βέβαια. Πάντως, Εντελώς συνοπτικά να πω ότι είναι 25% ο φόρος στις Ηνωμένε Πολιτείες, ενώ υπάρχει πιο χαμηλή φορολογική επιβάρυνση στην Ευρώπη. Πάντως και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού το θέμα της απλοποίησης των φορολογικών μέτρων είναι κάτι το οποίο θα μας άρεσε. Μιας και μιλάμε πολύ συχνά για το Λουξεμβούργο, να πω ότι εμείς το κεντρική έδρα μας στην Ευρώπη είναι στο Λουξεμβούργο. Έχουμε άνω των χιλίων ε, υπαλλήλων. Η ηγετική ομάδα της Amazon για την Ευρώπη είναι στο Λουξεμβούργο. Έχουμε επίσης ε, στις Βρυξέλλες ένα μικρό γραφείο λόμπι το οποίο αποτελείται από πέντε άτομα μόνο ε, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να μην υπάρξουν εμπόδια στην ψηφιακή αγορά γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκπρόσωπος του Facebook. Ε, σχετικά με τα BEPS πάντα, νομίζω ότι πολλά θέματα έχουν ήδη να αναφερθεί και μπορούμε να συμφωνήσουμε το Διεθνές Φόρουμ, δηλαδή αναφέρομαι στον ΟΣΑ, νομίζω ότι αυτό το οποίο ε, μπορεί να βοηθήσει είναι το ότι βασικός στόχος είναι η δημιουργία μιας σειράς διαλειτουργικών εναρμονισμένων κανόνων. Ο ΣΑ λοιπόν αποτελεί το φόρουμ για να το πετύχουμε. Να υπογραμμίσω επίσης τα πάρα πολύ υψηλά κέρδη που μπορεί να έχει κανείς από τις εργασίες που έχουν ξεκινήσει γύρω από τα BEPS. Νομίζω ακόμα και σε παιδαγωγικό επίπεδο μπορούμε όλοι να κερδίσουμε. Η προσπάθεια εξ αρχής είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Νομίζω ότι σήμερα είμαστε όλοι πιο ενήμεροι για τα θέματα αυτά και αυτό είναι θετικό στοιχείο. Για τα υπόλοιπα, τα όσα μπορούμε ακόμα να βελτιώσουμε, για το BEPS, εγώ δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ακούμε ότι ε, πρέπει ακόμα να ρυθμιστούν πολλές ε, λεπτομέρειες ε, για τους ορισμούς, για τις τιμελογήσεις, για τις μόνιμες έδρες και θα πρέπει λοιπόν να ρυθμιστούν αυτά, γιατί ε, ε, αλλιώ θα πέσουμε πάλι σε νομική ασάφεια, όπως ακούστηκε προηγουμένως. Και ενδεχομένως να υπάρξουν και ε, διαφορές, disputes όπως το λένε αυτό στα αγγλικά. για την επίλυση των διαφορών λοιπόν και των διεθνών συγκρούσεων μεταξύ των εταιριών. Έχει σημασία αυτό Πάντως καλώς ορίζουμε τις εργασίες που γίνονται ε, για αυτό το θέμα. Για το CCTB, τον ενιαίο, την ενιαία βάση φορολόγησης των επιχειρήσεων, ε, συμφωνώ. Έρχομαι τώρα στην ερώτηση της κυρίας Φερέρα και σας απαντώ κυρία μου για το τι συμβαίνει στην Αγγλία. Τι συνέβη συγκεκριμένα το 2014. Αυξήθηκε πώς να το πω τώρα, ε, ο αριθμός των εργαζομένων μας σε πολύ ψηλό βαθμό, οι οποίοι ε, αμείβονται με stock options. Ε, είναι πολύ σημαντικά λοιπόν όλα αυτά και οι ίδιοι εκφράζουν ικανοποίηση για το γεγονός ότι αμείβονται με stock options. Όλα αυτά ισχύουν για το 2014 και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, για τις κάτω χώρες. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ούτε Dutch sandwich, ούτε τίποτα τέτοιες ιστορίες, κατασκευάσματα για φορολογικά θέματα. Για το Λουξεμβούργο με ρωτήσατε τι κάνει το νομικό τμήμα. Το νομικό τμήμα ε, υποστήριξε μία ενδο ομιλική δανειοδότηση. Απλώς να πω για το Λουξεμβούργο το εξής. Για ποιο λόγο έγινε αυτό στο δίκαιο του Λουξεμβούργου. Διότι... Αυτό έχει να κάνει με τις διεθνείς συμβάσεις που διέπονται από το δίκαιο του Λουξεμβούργου και έχουν πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και σαφήνεια. Γι' αυτό επιλέγουν οι εταιρείε. Δεν πρόκειται ε, για καμία φορολογική προνομιακή μεταχείριση ή ευνοϊκή μεταχείριση στο Λουξεμβούργο σε καμία περίπτωση. Η κυρία Φερέιρα, μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι το γραφείο στις κάτω χώρες που έχετε δεν είναι μια θύρα ανοιχτή προς τους φορολογικούς παραδείσους. Αυτό το διαψεύδεται. Α, είναι εμπορικό το τμήμα εκεί, το γραφείο. Άρα ε, εμπορικό και τι πουλάτε. Ε, ε, παρακολουθούμε είναι ε, το μάρκετινγκ και τους μεγάλους λογαριασμούς. Και τα λεφτά που πάνε στα νησιά Καϊμάν από πού περνάνε. Μα εσείς τι ρωτάτε. Αν υπάρχει Dutch sandwich, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, Ολλανδικό sandwich. Δηλαδή δεν είναι ε, ένας τρόπος να μεταφέρονται. Ε, μα πώς πηγαίνουν τα λεφτά στα νησιά Κάιμαν, πετάνε. Ε, δεν ξέρω πώς να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Πάντω όχι μέσω των κάτω χωρών. Α, είναι μυστικό, λέει η κυρία Φεραίρα. Δεν είναι μυστικό, να απαντήσω ό,τι θέλετε. Μα σα ρωτάω και δεν μου απαντάτε αυτό που σα ρωτάω. Με χαρά να απαντήσω, απλώ δεν θέλω να σας παραπλανήσω λέγοντας κάτι που δεν ισχύει. Κατάλαβατε. Λοιπόν, μου έγινε και μια ερώτηση για ε, το συντελεστή που πληρώνει το Facebook στο FCC Filing στις Ηνωμένες ε, ε, πολιτείες, 40% για το 2014 και μου λένε αυτό πως υπολογίζεται ε, βάσει των ισχυών των κανόνων για το SSE filing. Αυτά είναι θέματα ε, λογιστικά. Αν θέλετε να μπω και σε λεπτομέρειες θα μπορώ να σας τα στείλω κιόλας. Γενικά, απαντώ για το lobbying, για την άσκηση πίεσης μια γενική ερώτηση που έγινε προς όλους, υποθέτω. Βεβαίως, στη διάθεσή σας για να απαντήσω. Κάνουμε και εμείς λόμπι. Ε, Ευρώπη, Ηνωμένε Πολιτείε, με διαφάνεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Λούντλαντ. Thank you very much. Um, Ευχαριστώ πολύ. Για τη διαδικασία Μπέψη, ήδη έχουν υποθεί πολλά. Απλώς να τονίσω ότι στη δικασία BEPS η ανάλυση που θα κάνουμε για το πού βρισκόμαστε στη διεθνή φορολογία είναι πολύ σημαντική. Όλα ξεκίνησαν πριν από μία διετία με μια πολύ μεγάλη στήριξη από τον ΠΕΠΣ γιατί θέλαμε μια διαφανή και ισότιμη φορολογική νομοθεσία και νομίζω ότι βοηθήσαμε να προχωρήσουμε όμως από το στόχο. Απλώ πρέπει να δούμε αν θα μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε κιόλα. Αυτό είναι το άλλο σκέλο τη ερώτηση. Δηλαδή, τι είναι πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή και νομίζω το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι συντονισμό σε όλη την Ευρώπη και με τι υπόλοιπε χώρε και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των κανόνων, των κανόνων BEPS, θα είναι πολύ σημαντικό τι 600 σελίδε γράφου που έχουμε στα χέρια μα να δούμε ακριβώ τι λεπτομέρειε πώ θα τι εφαρμόσουμε. Αυτό θα είναι το σωστό βήμα για να προχωρήσουμε. Για την Βερμούδα. Είναι το, η τρίτη πηγή φόρου για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί θα έπρεπε να φορολογούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μικρόφωνο. Είναι αγενές λέει ο μιλητής να σας γυρνάω την πλάτη. Αλλά εάν επαναπατρίζονταν τα εισόδηματα αυτά δεν θα φορολογούνταν. Θα έμεναν για επενδύσεις ή για άλλους σκοπούς αν επαναπατρίζονταν και φορολογούνταν, θα υπήρχε διαφορετική αξία. Δεν παράγεται όμω η αξία στι Βερμούδε. Ναι, όμω για όσα κάνετε στην Ιρλανδία και την Ολλανδία. Εκεί παράγεται αξία. Πού τα δηλώνετε, Στην holding τη Ιρλανδία. Και εκεί επισχύουν οι κανόνε τη ενιαία αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή γίνονται απολύτως σεβαστοί ε, όλοι οι κανόνες στις δηλώσεις των ε, εισοδημάτων σας. Ναι, μπορούμε να τα δώσουμε κιόλα και όπως είπα και στον ε, Πρόεδρο, μπορούμε να δώσουμε μια καταλεπτός παρουσιασμένη ανάλυση. Μέχρι εδώ φτάνουν βέβαια οι ερμοδότητέ μου, ε, για να σα τα εξηγήσω. Η τρίτη ερώτηση ήταν για τα φορολογικά συστήματα. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να συγκρίνουμε το αμερικανικό και το ευρωπαϊκό φορολογικό σύστημα, γιατί βασίζονται σε διαφορετικέ αρχέ. Κοιτάζουμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο και προσπαθούμε να βρούμε ποιο είναι ο σωστό τρόπο να το κάνουμε, να ακολουθούμε του κανόνε των φορολογικών συστημάτων με έναν συντελεστή 19,3% συνήθως και το 80% να πληρώνεται στις ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή έτσι ε, έχει οργανωθεί το φορολογικό σύστημα και έτσι εφαρμόζεται. Αυτό που θα ήθελα να πω εν τέλει είναι ότι συμμετέχουμε σε διάλογο και συζητήσεις με τον ΩΣΑ και με όλους τους υπόλοιπου που θέλουν να συζητήσουμε για το φορολογικό σύστημα και πώ θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο. Και βεβαίω και θα μπορούσε αυτό να ονομαστεί lobbying, αλλά αυτή η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί πιστεύω, γιατί θα πρέπει να είναι κανόνε προβλέψιμοι, σαφεί, διαφανεί και να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση σε καμία περίπτωση. Να μπορούμε να του δούμε και να του εφαρμόσουμε. μια ε, διευκρινιστική ερώτηση. Δηλαδή, όσα πάνε στην Βερμούδα δεν φορολογούνται πουθενά. Στι Βερμούδε λοιπόν δεν φορολογούνται ποτέ, ποτέ ε, από το 19% των ΗΠΑ ε, πηγαίνουν προς τις Βερμούδες για να επενδυθούν αλλού, δεν φορολογούνται. Δεν μπορώ να σας πω αν θα φορολογούνταν εφόσον επαναπατρίζονταν τα ποσά αυτά. Ε, ναι, αλλά ακριβώ μετακινούνται για να μην φορολογηθούν. Ναι, πηγαίνουν σε ξένες επενδύσεις. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, μια σύντομη διευκρίνηση. Ευχαριστώ. Μια σύντομη διευκρίνηση. Αναφέρατε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε μπορούν να επηρεάσουν και όχι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννοείται την Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμό ή εννοείται τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωση. Τι εννοείται να επηρεάσουν. Με συγχωρείτε. Με τους φόρους που φεύγουν από τι ΗΠΑ. Λέτε ότι δεν υπάρχει αντίκτυπο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννοείται την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά ω ε, θεσμό, ω οργανισμό ή εννοείται τα κράτη-μέλη. Του τους φόρους που θα καταβάλλονταν στα κράτη-μέλη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε στο σύστημά του, έχουν την αρχή του deferral. Δηλαδή τα κέρδη εκτό Αμερικανική επικράτεια δεν φορολογούνται ευθύ αμέσω. Υπάρχει ετεροχρονισμένη φορολογία. Ίσως τον 22ο-23ο αιώνα να είναι η αναβολή. Αλλά υπήρξε η αλλαγή αυτή με την κυβέρνηση Κέννεντι που την επανέλαβε ω νόμο και η κυβέρνηση Ρίγκαν. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους παρεμβαίνοντες συμπληρωματικά να πω ότι θα χρειαστούμε ένα κείμενο της Google που να εξηγεί, να δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις που τόσο πολύ, στις οποίες τόσο πολύ επεκταθήκαμε για το Double Irish και το Ολλανδικό sandwich το οποίο το τρώνε και ο Αμερικανός και ο Ευρωπαίος φορολογούμενος τελικός και κατά τα άλλα για τις αμοιβέ, για όσα δηλαδή λαμβάνει το Φορολογικό Συμβούλιο, το Facebook, η εκπρόσωπος του Facebook επιβεβαιώνει είπαμε, κυρία μου, σωστά, ότι δεν είναι ανάλογη, ανάλογα τα ποσά που καταβάλλονται με το φόρο που έχει αποφευθεί, από τον οποίο υπήρξε έκδοση. Και από την άλλη, κυρία Ζολή θα ήθελε το σύνολο των επιχειρήσεων που εκπροσωπούνται σήμερα εδώ να μας ε, σημειώσουν το κόστος των φορολογικών συμβούλων το σύνολο των αμοιβών που καταβάλουν προς ε, την συμβουλευτική για τις επιχειρήσεις ιδίω που έχουν εκθέσεις χώρα, είναι εύκολο να δώσουν αυτά τα στοιχεία. Οι υπόλοιποι θα έπρεπε ίσως λίγο να ψάξουν, αλλά θα θέλαμε να έχουμε απαντήσεις ως το τέλος της εβδομάδας, γνωρίζοντας ότι οι απαντήσεις αυτές μπορεί να αποσταλούνται με email, δηλαδή μέσω Google, είτε με δέμα από την Amazon, είτε με τα κοινωνικά δίκτυα μέσω Facebook. Σας ευχαριστώ και κάνουμε ένα λεπτό διακοπή για να φύγουν οι προσκεκλημένοι αυτού του πάνελ και να έρθουν αυτοί του επόμενου.